Ladies uh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ο πρόεδρος ε, κύριος Τραγάκης ε, και εγώ θα ξεκινήσουμε την ε, επόμενη συνεδρία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας εξηγήσω για μια ακόμη φορά ότι έχουμε δίλεπτες παρεμβάσεις τους ομιλητές, αλλά και μια εισαγωγική ομιλία από τον Επίτροπο Όλη Ρέν, προκειμένου τον οποίο θέλω να καλωσορίσω για μια ακόμη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι σε καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά εδώ. Μετά λοιπόν την ομιλία του Όλη Ρέν θα έχετε οι συνάδελφοι 4-5 τον αριθμό, το λόγο για δύο λεπτά ο καθένας. Θα ακούσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έναν ε, συνάδελφο. Ο κύριος Τράκης και εγώ, όπως είπα, συμπροεδρεύουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Όλη Ρέν, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις οικονομικές νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ αν θέλετε, είναι ο Υπουργό Οικονομικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Επίτροπε, αγαπητέ Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Thank you. Thank you, Chair. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αγαπητέ Ότομάδα. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ των Εθνικών Κοινοβουλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτον, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση να μετάσχω στην κοινοβουλευτική στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα και στην διάσκεψη που οργανώνεται για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ε, θεσπίζεται από τη συνθήκη για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Η διάσκεψη νομίζω ότι είναι μια σημαντική συμβολή στην οικονομική διακυβέρνηση. Η δε συνάντησή μας αυτή μας δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές στην Ευρώπη και να ενισχύσουμε την νομιμοποίηση της διαμόρφωσης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πω δύο λόγια καταρχάς για την δημοσιονομική πολιτική που τυπικά τουλάχιστον βάσει της σημερινής διάταξης που έχουμε είναι στο κέντρο των σημερινών συζητήσεων. Και κατόπιν θα πω και λίγα λόγια για την οικονομική κατάσταση και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις χώρες της Ευρωζώνης. Ξεκινώ με τα δημοσιονομικά θέματα. Οι ρίζες της κρίσης βρίσκονται και σε δημοσιονομικές και σε μακροοικονομικές ανισορροπίες που διαμορφώθηκαν την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της κρίσης έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά μέτωπο για να αποφύγουμε χειρότερα σενάρια και να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη. Μετά τα αρχικά δημοσιονομικά μέτρα παρέμβασης που συντόνισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αποκατάστασης όπως λέγεται μεταξύ του 2008 και 2009, η Ένωση χρειάστηκε να αναλάβει μια, ένα φιλόδοξο καθήκον για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την υγεία των δημοσίων οικονομικών. Η κοινή αυτή στρατηγική βασίστηκε σε τρεις ε, βασικές καθηγητήριες γραμμές. Πρώτον, διαφοροποίηση, δηλαδή το μέγεθο και ο επίγον χαρακτήρα των δημοσιονομικών προκλήσεων ποικίλουν από κράτο σε κράτο. Κατά συνέπεια, ε, ο βαθμό και η ταχύτητα εξυγίανση ήταν διαφορετικέ. Οι χώρε που είχαν μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο και λιγότερη πίεση να κάνουν front-loading στην εξυγίανση από ότι άλλε χώρε με μικρότερο δημοσιονομικό περιθώριο. Δεύτερον, τονίζουμε, τονίζαμε εξ αρχή ότι η επιλογή των μέτρων εξυγίανση θα έπρεπε να λάβει η υπόψη τα αποτελέσματα των μέτρων ανάπτυξης, των αναπτυξιακών μέτρων και τα μέτρα που μείωναν, που ε, ήταν λιγότερο επιβραβείς για την, για την ανάπτυξη θα πρέπει να λάβουν ε, πιο μεγάλη προτεραιότητα. Καταλαβαίνω ότι κάποιες χώρες χρειάστηκε να κάνουν δύσκολες επιλογές. Είμαι ωστόσο πεπισμένος ότι η έλλειψη εξυγένσης σε τέτοιες περιπτώσεις θα είχε οδηγήσει σε ακόμα χειρότερες συνθήκες, ιδίως αν ε, είχαν κλείσει τι πόρτε τους οι οικονομικές αγορές στι χώρε αυτές, όπως συνέβη σε ορισμένα κράτη-μέλη. Τρίτον, οι προσπάθειες ε, της δημοσιονομικής εξυγίανσης θα έπρεπε να συνοδεύονται και να υποστηρίζονται από διαφορετικέ μεταρρυθμίσει για τη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξη μέσω πρόθεσμα και να καταστήσουν ε, να δώσουν βιώσιμα αποτελέσματα στην εξυγίανση. Σήμερα, παρότι θα έπρεπε να αποφύγουμε οποιαδήποτε ε, έκφραση ικανοποίηση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η συνολοποιημένη δημοσιονομική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σταδιακά μετατρέπεται σε βιώσιμη. Οι σημαντικές προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια δίνουν τώρα αποτελέσματα σε αυτό το τρίμηνο. Δύο παρατηρήσεις. Το ονομαστικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2014 φέτος αναμένεται να πέσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ για πρώτη φορά στην πράξη από το 2009. Αυτό δεν είναι μόνο προβολή, αλλά εδράζεται και σε σχέδια προπολογισμό που εσείς εγκρίνατε και, και εσείς ως κράτη-μέλη στηρίζονται λοιπόν σε συγκεκριμένες αποφάσεις πολιτικής από τις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια. Δεύτερον, το επίπεδο του δημοσίου χρέους αναμένεται φέτος να σταθεροποιηθεί γύρω στο 90% του ενωσιακού ΑΕΠ Όταν ξεκίνησε η κρίση, το, ε, χρέος στην Ευρώπη ήταν συνολικά 60% ε, του ΑΕΠ. Το αποτέλεσμα της κρίσης ήταν η αύξηση κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες στο 90%. Αλλά σταθεροποιήθηκε και αυτό είναι καλά νέα από την οπτική γωνία των βιώσιμων δημοσίων οικονομικών. Τα αποτελέσματα είναι ότι οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι μειώθηκαν όσο ενώ ο βαθμός εξυγίανσης μετριαζόταν, θα μπορούσε να μετριαστεί. Και τούτο αντικατοπτρίστηκε στις αποφάσεις που λήφθηκαν πέρυσι το φθινόπωρο και, ε, την άνοιξη και το καλοκαίρι. Όταν το Συμβούλιο βάσει συστάσεων της Επιτροπής επέκτηνε κάποιες ε, προθεσμίες διόρθωσης των υπερβολικών ελλημάτων εν και των προσπαθειών των κρατών μελών και των τότε αντίξεων οικονομικών συνθήκων σε κάποια κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα την Ισπανία και την Πορτογαλία ή σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για διαφορετικές μεταρρυθμίσεις στην Γαλλία, την Ολλανδία και κάποια άλλα κράτη-μέλη. Ωστόσο, η σε οτι αφορα τις δεσμευσει για διαφορετικες μεταρρυθμισεις αυτή κρατη ωστοσο η γενικη αυτη εικονα κρύβει σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχουν χώρες όπου οι δημοσιονομικές ανισορροπίες απαιτούν μεγαλύτερη ενίσχυση των δημοσιονομικών θέσεων. Αγαπητοί φίλοι, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση συνολικά στην Ευρώπη, θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για την συζήτησή σας ξεκινώ μιλώντας για την Ελλάδα, διότι είναι και η ελληνική προεδρία. Έχουμε ελληνικό, Έλληνα συμπρόεδρο στην συνεδρίαση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισκέφθηκε πριν από δύο εβδομάδες ε, την ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα ε, στο ξεκίνημα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ένωσης. Τότε υπήρχαν ενθαρρυντικά οικονομικά νέα που συνέπεσαν με ένα πολύ ωραίο λαμπερό καιρό, λαμπερό ουρανό στην Αθήνα. Τώρα, στη συνάντηση, μάθαμε ότι ο δείκτης οικονομικών, ε, ε οικονομικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε συνολικά σε για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2011. Η, η άνοδος αυτή του δείκτη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι ισχύει και για τις ε, τροτές χώρες. Μεταξύ δε αυτών υπάρχει και ο δείκτης ε, εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Και αυτό συνοδεύεται και από σταθερά στοιχεία για, την, για το λιανεμπόριο, ενώ και, την εικόνα ότι η αγορά εργασίας σταθεροποιείται. Ο, πρόσφα, πιο πρόσφατος δείκτης έρευνας ε, αγοραστικής ικανότητας υποστηρίζει την θέση μας για μια μικρή δημοσιονομική ε, ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους στην Ευρώπη. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι τα θετικά νέα έρχονται εκτός Γερμανίας. Υπάρχουν δηλαδή θετικά νέα και από αλλού. Χώρες που πριν ή συνεχίζουν ακόμα για λίγο διάστημα να υπάρχουν σε προγράμματα αναδιάρθρωσης. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, που θα βγει από το πρόγραμμα σταθεροποίησης σε 34 ώρες περίπου από τώρα. 32 ώρες διορθώνει ο μιλητής. Διότι λύγει το πρόγραμμα τα μεσάνυχτα της 22 Ιανουαρίου. Ο τραπεζικός κλάδος της Ισπανίας επισκευάστηκε και, οι σημαντικές ε, οικονομικές μεταρρυθμίσεις ε, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Τα, οικονομι... τα αισθήματα για την οικονομία επανήλθε στο μακροπρόθεσμο μέσο όρο για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2007. Επιπλέον, η Ιρλανδία επανήλθε πριν από δύο εβδομάδες περίπου στις αγορές για πρώτη φορά μετά τη σύναψη του προγράμματος τον Δεκέμβριο με πολύ χαμηλότοκα δεκαετή ομόλογα. Το πρόγραμμα ξεπερνά το 7% το Νοέμβριο του 2010 και κάποια στιγμή είχε φτάσει, είχαν φτάσει τα επιτόκια στο 14%. Τα πράγματα άλλαξαν πολύ σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια για την Ιρλανδία. Βλέπουμε λοιπόν φρέσκα βλαστάρια, αλλά ο τραπεζικός τομέας συνεχίζει να έχει κάποια αβεβαιότητα. Η, οικονομία της Ευρώπης συνεχίζει να αντιμετωπίζει ανάγκες διαθροτικών αλλαγών και είναι σημαντικό το χρηματοοικονομικό σύστημα να παράσχει πόρους στις πιο δραστήριες και χρήσιμες χρήσεις. Είναι σαφές ότι για πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πολίτες της Ένωσης η εποχή συνεχίζει να είναι δύσκολη, καθότι η ανεργία παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες απαιτούνται, συνεχίζουν να απαιτούνται συνεχιζόμενες προσπάθειες για την βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, παράλληλα με τις ε, συνεχιζόμενες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και την ενίσχυση του, των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων η στρατηγική διαθροτικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να πηγαίνει με υγιή δημοσιονομική, ε, κρατική δημοσιονομική πολιτική και θα δώσει σύντομα ε, και θα δώσει γρήγορα θετικά αποτελέσματα. Το είχε δείξει αυτό και η περίπτωση της Λετωνίας. Πριν από λίγο καιρό επισκέφθηκα την ε, Λετωνία για να καλωσορίζω το 18ο μέλο της ζώνης του ευρώ. Πριν από δύο χρόνια η Λετωνία πέρασε μια τρομερά βαριά ύφεση, είχε, είχε στηριχθεί με προγράμματα του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, τώρα όμως είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της Ένωσης. Οι Κασάνδρες λοιπόν διαψεύστηκαν. Η στρατηγική που επέλεξε η Ευρώπη για να ξεπεράσει την κρίση δουλεύει. Και η στρατηγική ακολούθησε την προσέγγιση της επέκτασης της αλληλεγγύης για σε αντάλλαγμα με σταθερότητα. Αυτό, απαιτεί, αυτό ε, απαιτούσε δεσμεύσεις, σοβαρές δεσμεύσεις των κρατών μελών που λάμβαναν ενίσχυση για να αντιμετωπίσουν τις συσσωρευμένες ανισορροπίες τους, να εφαρμόσουν ε, μεταρρυθμίσεις και να αναμορφώσουν την δημοσιονομική τους ε, κατάσταση σε βιώσιμο επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, σε αυτό το σταυροδρόμι μπροστά σε μια οικονομική ανάπτυξη που ανάκαμψη που ξεκινά, είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε στην πορεία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων για να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και κυρίως για, τη... για τις μελλοντικέ γενιές. Η εμπιστοσύνη επανέρχεται. Τούτο τόσο δεν σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να κινδυνεύσουμε να χάσουμε το momentum των μεταρρυθμίσεων αντί να εξυγχρονίσουμε και να μεταρρυθμίσουμε τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας για να ενισχύσουμε την ικανότητα ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και αντιμετώπισης άλλων προκλήσεων. Πιστεύω ότι το τεστ αυτό θα το ξεπεράσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Περιμένω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την εισαγωγή σας. Προχωράμε στη συζήτηση. Να δώσω το λόγο στον πρώτο ομιλητή, κύριο Παπαδημούλη από την Ελλάδα. Κύριε Επίτροπε, εσείς παρουσιάζοντας το παράδειγμα της Ελλάδας με κάποια στοιχεία, είδατε φρέσκα βλαστάρια. Εγώ σας μεταφέρω μια τεράστια οικονομική και κοινωνική καταστροφή που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν μεγάλες ευθύνες για το πώς φτάσαμε εκεί με ελλείμματα, με χρέη, με γραφειοκρατία, με διαφθορά. Αλλά το δικό σας μνημόνιο προέβλεπε συνολική ύφεση 14% και ήδη έχουμε φτάσει στο 25. Προέβλεπε το πικ της ανεργίας 14% και έχουμε φτάσει στο 28. Προέβλεπε ότι θα αρχίσει να μειώνεται το δημόσιο χρέος και πριν μπούμε στα μνημόνια ήταν 125% και τώρα είναι 175%. Και έχουμε και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Και οι υγιείς επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στην τραπεζική ρευστότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο βλέπει έλλειμμα δημοκρατίας διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας στο πώς λειτουργεί η τρόικα και στην ελλάδα και στις άλλες χώρες. ποια είναι η δική σας γνώμη; όλα καλά; εσείς παραδεχθήκατε ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε όλη την ευρωζώνη από το 60% στο 90%. Ποια είναι η γνώμη σας για μια πρόταση που κερδίζει διαρκώς έδαφος που ζητά ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος για να δοθεί ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό και όχι μόνο ευρωπαϊκή απάντηση στο θέμα των τραπεζών. Μιλήσατε πάνω από δέκα λεπτά. Δεν αναφέρατε μια φορά τη λέξη συνοχή. Και όμως στις πολιτικές της κοινότητας και στη της Λισαβόνας μιλάνε τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολιτική συνοχής εδαφικής, κοινωνικής, περιφερειακής σας ερωτώ, είναι τυχαία αυτή η παράληψη στην ομιλία σας και πώς μπορούν να υλοποιηθούν πολιτικές συνοχής που να μειώνουν τις εκρηκτικές ανισότητες κοινωνικές, εδαφικές, περιφερειακές όταν η Κομισιόν και το Συμβούλιο συνομολογούν προϋπολογισμό ευρωπαϊκό λιγότερο από το 1% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου προϊόντος. Και τέλος, επειδή έχετε έναν τόνο εφορίας και κατηγορείτε τις Κασάνδρες που είναι αρχαία ελληνική παράδοση. Μπορείτε να μου πείτε γιατί η Ευρωζώνη με τις δικές σας συνταγές τα πηγαίνει πολύ χειρότερα από την Αμερικανική οικονομία που εφαρμόζει πιο κενσιανές μεθόδους. Και στο κάτω-κάτω της γραφής η κρίση ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Our next Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφός μας από την Βουλή των Λόρδων, ο κύριος Χάρισον. Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ρεν που συναντήθηκε με την Επιτροπή μου για την ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση τον Οκτώβριο. Θα μπορούσε να μου απαντήσει στις εξής ερωτήσεις. Καταρχάς, εάν η Τραπεζική Ένωση είναι κεντρική. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα εγγύησης καταθέσεων ή άλλα προγράμματα είναι λιγότερο κεντρικά. Και όσον αφορά τον ε, μηχανισμό ε, ανάκαμψης των τραπεζών, πιστεύετε ότι υπάρχουν αρκετά χρήματα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαβούλευση 200 ε, ανθρώπων ε, ή οργανισμών μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και ποιες πιστεύετε ότι είναι οι συνέπειες για τις 10 χώρες που δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη. Κάποιες από αυτές θέλουν να προσχωρήσουν, άλλες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να μην προσχωρήσουν σύντομα. Και τέλος, Πότε πιστεύετε ότι θα έχει ξεπεραστεί η κρίση, πώς θα γνωρίζουμε ότι έχει ξημερώσει η ημέρα που μπορούμε να επανέλθουμε στις κανονικές μας δουλειές, πώς θα γνωρίζουμε ότι έχουμε επιλύσει την κρίση που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία 6-7 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σούτ είναι η συγητής ε, του Κοινοβουλίου των Κάτω Χωρών για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Συγγνώμη, κυρία. Κύριε Πρόεδρε. Σας μιλώ ως εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο της Βουλής Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω εσάς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που, που οργανώσατε αυτήν την διακοινοβουλευτική διάσκεψη. Χαίρομαι που έχουμε αυτή την ευκαιρία να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική ύφεση στην Ευρώπη η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου είναι υπέρ του συντονισμού των ε, δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών ώστε να ε, μπορέσουν να περάσουν στην ευημερία οι οικονομίες. Η πολιτική των κρατών μελών όχι μόνο συμβάλλει σε ένα κοινό στόχο με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ο συντονισμός δεν αφορά μόνο τις χώρες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Οι εξαγωγικέ αγορές όλων των κρατών μελών σχετίζονται μεταξύ τους, έτσι θα υποφεληθούμε όλοι από την καλύτερη συνεργασία. Καταρχάς θα ήθελα να συνοψίσω τις ε, μεταρρυθμίσει του 2014 και να εξετάσω τι ε, προτεραιότητε του 2014. 8 τρίμηνα ύφεση ε, έχουν επηρεάσει τις κάτω χώρες. Ε, το διαθέσιμο εισόδημα δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το 2013 ήταν γνωστό για την αύξηση της ανεργίας ε, και τον υψηλό πληθωρισμό. Οι κάτω χώρες έπρεπε να αντιμετωπίσουν ασταθείς κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες λόγω των μεταρρυθμίσεων. Και το 2013 έχει υπάρξει μεγαλύτερη διάθεση για μεταρρυθμίσεις. Θα είναι λιγότερο αυστηρή η κοινωνική προστασία για τους ε, ανέργους, θα δοθούν όμως περισσότερες ε, θέσεις εργασίας ε, στους αναπήρους. Όσον αφορά την κοινωνική στέγαση, τα ενίκια βρίσκονται στο μέγιστο ε, αλλά θα μπορούν να γίνουν ε, ε, αυξομοιώσεις ανάλογα με το εισόδημα των κατοίκων. Επίσης θα μειωθούν κάποιοι φορολογικοί συντελεστές. Έχουμε και μεταρρυθμίσεις στην υγεία και στις συντάξεις, αλλά θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι οι κάτω χώρες ε, έχουν αφιερώσει μέρος ε, του προϋπολογισμού ε, στις μεταρρυθμίσεις αυτές. Έτσι λοιπόν οι Υπουργοί πρέπει να εξηγήσουν πώς εφαρμόζουν τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέρφους να συνομιλήσουν και να μάθουν ένας από τον άλλον τώρα στις εποχές αυτής της κρίσης. Θα ήθελα να γνωρίζω εσείς πώς βλέπετε τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Σαχινίδης από την Ελλάδα. Παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Ρέν για την παρέμβασή του. Η παρέμβασή μου αφορά την αλληλεπίδραση δημοσιονομικής προσαρμογής και αναπτυξιακής προοπτικής και απασχόλησης των χωρών που είναι σε οικονομικό πρόγραμμα η Ελλάδα το 2013 συμπληρώνει έξι χρόνια ύφεση έχοντας χάσει πάνω από το 1 τέταρτο του εθνικού εισοδήματος. Είναι η μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος στη σύγχρονη ιστορία, μεγαλύτερη και από αυτή που είχαν οι Ηνωμένε Πολιτείες μετά την κρίση του 1929. Όσοι παρακολουθούν την πορεία προσαρμογής της Ελλάδος τονίζουν την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιστρέψει η Ελλάδα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι σωστό ότι η Ελλάδα πριν ξεσπάσει ακόμα η κρίση χρειαζόταν να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών και εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις όμως από μόνες τους δεν βοηθούν την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα αλλά μόνο μέσω μακροπρόθεσμα. Σήμερα όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι το πρόβλημα της χώρας είναι πλέον πρόβλημα ζήτησης και όχι προσφοράς. Η δημοσιονομική πολιτική στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι συσταλτική στα επόμενα χρόνια ώστε να πετύχει το στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα και να θέσει σε έλεγχο τη δυναμική του χρέους. Αρνητική ή μηδενική συνεισφορά στη ζήτηση θα έχουν και η κατανάλωση λόγω της υψηλής φορολογίας της μείωσης των εισοδημάτων αλλά και της ανεργίας αλλά και οι επενδύσεις αφού οι περισσότερες επιχειρήσεις δουλεύουν στο 60% της δυναμικότητάς τους. Την ίδια στιγμή όλες οι ελπίδες για την ανάπτυξη έχουν στηριχθεί στις καθαρές εξαγωγές είναι γεγονός ότι οι εισαγωγές μειώνονται αλλά δεν υποκαθίστανται από εγχώρια παραγωγή. Οι εξαγωγές εμφανίζουν σημάδια κόπωσης. Με βάση τα προαναφερθέντα, από πού πιστεύετε ότι θα έρθει η ανάπτυξη στην Ελλάδα στα επόμενα χρόνια αφού πλέον είναι πρόβλημα ζήτησης και όχι προσφοράς. Ευχαριστώ. Mr. Popak. Yeah, you, but you are not. No. So, Herr Kommissar, bitte. Κύριε Πίτροβε, παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, βουλευτές ε, για τα πολύ ουσιαστικά ερωτήματα που έθεσαν. Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό οι παρεμβάσεις ε, περίχαν και πολιτικά σχόλια, όχι τόσο ερωτήσεις. Τα θέματα πάντως τα οποία ετέθησαν, που ήταν ερωτήσεις πιο πολύ, θα προσπαθήσω να τα απαντήσω. Καταρχάς, ό,τι αφορά την παρέμβαση του κυρίου Παπαδημούλη για το ελληνικό πρόγραμμα. Έχετε μια σταθερή ε, γραμμή και με τον ε, σύντροφό σας τον κύριο Χουντή διότι τον ακούω πάντοτε στην ε, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου και πάντοτε εκφράζει την ίδια κριτική κατά της Κομισιόν και κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα τελευταία χρόνια ακούω ε, τις κριτικές για το Διεθνούς Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να σας πω ότι η απόφαση τη Ευρωζώνη, η απόφαση τη Κομισιόν να στηρίξει την Ελλάδα δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά ήταν μια υπεύθυνη απόφαση. Διότι αν αφήναμε την Ελλάδα χωρίς διάσωση οικονομική πριν από τέσσερα χρόνια το 2010, η Ελλάδα θα είχε πέσει και μάλιστα με ελεύθερη πτώση και θα είχαμε οικονομική καταστροφή της χώρας και οι επιπτώσεις ε, θα μεταδίδονταν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η διάγνωση που κάναμε ήταν ότι το ελληνικό πρόγραμμα ξεκινά από ε, δημοσιονομική ανευθυνότητα, κάποια στατιστικά ε, προβλήματα, στατιστική απάτη θα έλεγα μάλιστα και προβλήματα ανταγωνιστικότητας μεταξύ άλλων τα οποία θεωρήσαμε ότι έπρεπε να διορθωθούν με διαρθρωτικά και δημοσιονομικά μέτρα. Οι δημοσιονομικοί στόχοι μετά από διάφορες δυσκολίες λίγο πολύ πλέον ε, επετεύθησαν, αλλά δυστυχώς καθυστέρησαν οικονομικές μεταρρυθμίσεις λόγω των συμφερόντων και λόγω της πολιτικής αντίδρασης και αντίστασης της κοινωνίας. Και αυτό έκανε να μην έχουμε ακόμη ανάκαμψη και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο μου γίνει αυτή η ανασκόπηση της ελληνικής κατάστασης και σε άλλους βουλευτές γιατί πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ξανασυζητήσουμε ε, τα θέματα της Ελλάδας και καλό θα ήταν όλοι να γνωρίζουν πού βρισκόμαστε. Πρέπει να σας πω ότι αναμένουμε σταδιακή επιστροφή στην ανάπτυξη από φέτος επειδή βελτιώνεται η οικονομική διάθεση, η εμπιστοσύνη και περιμένουμε και να έχουμε και επενδύσεις φέτος ο λόγος ε, χρέους ΑΕΠ αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται από του χρόνου και την επόμενη δεκαετία να πέσει κάτω από το 120%. Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρμογή του προγράμματος, οι ελληνικές αρχές καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες. Οι σταθμοί, τα ορόσημα που έχουν να κάνουν με την ε, ταμείευση ε, της τρίτης δόσης μετά την αξιολόγηση δηλαδή, ολοκληρώθηκαν τις σχετικές διαδικασίες στις 17 Δεκεμβρίου, αλλά πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά. Έχουμε την τέταρτη εξολόγηση. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται οι συνομιλίε ε, για μια σειρά πολιτικών που θα αποτελέσουν τη βάση επιτυχή ολοκλήρωση τη αξιολόγηση, τη τρέχουσα αξιολόγηση. Υπάρχει πρόοδο. Παραμένουν ωστόσο κάποια ανοιχτά ζητήματα για τα οποία απαιτείται μεγαλύτερη δουλειά, περισσότερη δουλειά και ελπίζω οι ομάδες ε, της αξιολόγησης να μπορέσουν να επανέλθουν στην Ελλάδα εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί βέβαια το έργο των ελληνικών αρχών σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες και τις δημοσιονομικές τους προσπάθειες. Με ρωτήσατε αν η Ελλάδα θα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα. Για πέρυσι ε, είδαμε ότι ήταν εφικτός αυτός ο στόχος. Και σίγουρα το πρωτογενέ πλεόνασμα αποτελεί προπόθεση για την αντιμετώπιση του ζητήματο τη βιωσιμότητα του χρέου. Κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε αργότερα, φέτο, η διάρκεια του τρέχοντο. Ε, πιο πολλά πρέπει να γίνουν, ιδίω σε ό,τι αφορά ε, τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματο ε, και τη ε, διαχείριση των εσόδων. Επίση και η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, τη δημόσια διοίκηση, είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημα του Λόρδου Χάρισον για το κοινό πρόγραμμα εγγύης των καταθέσεων. Η υπόθεσή σας ήταν σωστή. Δεν είναι για σήμερα, είναι για αύριο, για μεθαύριο. Τώρα εστιάζουμε στην υλοποίηση του ενίου εποπτικού μηχανισμού και την ε, οριστικοποίηση του ε, νέου ε, μηχανισμού εξυγίανσης των τραπεζών και τη συγκρότηση του σχετικού ταμείου εξυγίανσης. Η Κομισιόν θα επανέλθει πάντως αργότερα και σε αυτό το θέμα για ένα κοινό πρόγραμμα και σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Είπατε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τα κράτη μέλη που είναι εκτός Ευρωζώνης. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε πάντο δυνατόν στο πλαίσιο της ενίας αγοράς των 28 κρατών μελών της Ένωσης, συνολικά δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν κάποιες ειδικέ ανάγκες για την Ευρωζώνη ε, που πρέπει ε, να εμβαθύνουμε και στην δημοσιονομική κυριαρχία και στην ολοκλήρωση. Ο Τζόρτζ Όσμπορν, Υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε πει ότι το ενιαίο νόμισμα φέρνει μαζί του και την ανάγκη της βαθύτερη ολοκλήρωσης οικονομικής και δημοσιονομικής. Είναι μια φράση πλέον περιβόητη και είναι η αλήθεια ότι θα πρέπει να βαδίσει ε, ταχύτερα η Ευρωζώνη σε αυτό το μονοπάτι σε σχέση με τι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί για το ενιαίο νόμισμα απαιτείται και νομισματική αλλά και σταθερή εύρωστη οικονομική ένωση για να μπορέσει να στηριχθεί αυτό το νόμισμα. Πότε θα έχει ξεπεραστεί η κρίση, με ρωτήσατε. Κατά την άποψή μου θα έχουμε επανέλθει ε, σε ισχυρό ποσοστά, σταθερά ποσοστά ανάπτυξη και θα έχουμε αξιοποιήσει το δυναμικό μας το αναπτυξιακό ε, όταν θα έχουμε και ε, απασχόληση αύξηση της απασχόλησης. Στο σωστό δρόμο βρισκόμαστε. Είμαστε στο δρόμο της οικονομικής ανάκαμψης, η οποία είναι βιώσιμη, αλλά πρέπει αυτή την ανάκαμψη να την ενισχύσουμε και να ε, αξιοποιήσουμε όλο μας το δυναμικό για να επιταχυνθεί η δημιουργία απασχόλησης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Για την κυρία Σουτ από τις κατοχώρε, η οποία μας έκανε μια πολύ έτσι, χρήσιμη επισκόπηση της ε, οικονομικής και πολιτικής κατάστασης των κατοχωρών. Θέλω να πω λοιπόν στην κυρία Σούτσα ότι παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, τις συστάσεις τις οποίες διατύπωσε το Συμβούλιο προς τα κράτη-μέλη. Θα επανέλθουμε στη... στα θέματα αυτά την Άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού. Σε ό,τι αφορά στις χειμερινές προβλέψεις για κάποιες χώρες, αυτές θα επικαιροποιήσουν την οικονομική μας εκτίμηση γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε και τότε θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή μας για το κατά πόσον ε, είναι σε βιώσιμο δρόμο οι δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών. Μια πληρέστερη αξιολόγηση των οικονομικών και δημοσιομικών πολιτικών θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Οπότε και θα αξιολογήσουμε τόσο τις δημοσιονομικές πολιτικές όσο και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών. Για τον κύριο Σαχινίδη ο οποίος έθεσε ε, ένα ερώτημα για την Ελλάδα. Σας παραπέμπω και στην προηγούμενη απάντησή μου για τις εξελίξεις και για τις προσδοκίες που έχουμε για την Ελλάδα και την υλοποίηση του προγράμματος. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ραν για τις απαντήσεις. Το λόγο έχει ο κύριος Αντρέη Καζαλεύσκη, Καλαζεύσκη από το Πολωνικό Κοινοβούλιο. Mr. Kalazewski. No. Το λόγο έχει από την Ελλάδα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο κύριος Περμάστερ. Sorry, but uh, what? Wait. Is I will uh, have an intervention in the next uh, topic. Ε, συγγνώμη, έχω μια παρέμβαση για το επόμενο θέμα. για τη συζήτηση πάνω στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κρεμαστινός, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου ε, να ρωτήσω τον κύριο Όλιρε, ε, με τους Έλληνες συναδέλφους και για να μην επαναλάβω τα ίδια, με το θέμα των ελληνικών τραπεζών. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι έχει γίνει ένα haircut των ομολόγων στις τράπεζες. Είναι γνωστό ότι έχει γίνει επανακεφαλαιοποίηση και με τις δικές σας δηλώσεις είπατε ότι υπάρχει εγγύηση των καταθέσεων κάτω από 100.000 ευρώ. Ε, ότι οι ελληνικές τράπεζες καταθέτες κατά το 85 με 90% είναι καταθέτες κάτω των 100.000 ευρώ. Όμως έχουν φύγει οι μεγαλοκαταθέτες και σήμερα περί τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ βρίσκονται στις ε, τράπεζες της Κεντρικής Ευρώπης και στην Ελβετία. Οι τράπεζες είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να γίνει ανάπτυξη. Και πολύ φοβούμε ότι και οι καταθέτες των 100.000 ευρώ και κάτω θα αρχίσουν να σκέφτονται μήπως συμβεί το ίδιο πράγμα που συνέβη ενδεχομένω στην Κύπρο με μικρότερο, με, με μικρότερο αριθμό, δηλαδή λιγότερο από τα 100.000 ευρώ. Έχω την εντύπωση ότι με αυτόν τον τρόπο είναι αδύνατο να γίνει ανάπτυξη στην Ελλάδα όταν οι τράπεζες στην πράξη σήμερα δεν μπορούν να ενισχύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα κανένας δεν δανειοδοτείται πρακτικά στην Ελλάδα. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν, εάν δεν γίνει μια κατηγορηματική δήλωση ότι δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις, τουλάχιστον στις τράπεζες των χωρών που πρέπει να γίνει ανάπτυξη, πώς είναι δυνατόν το πρόγραμμα αυτό να προχωρήσει και πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη για να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα που οι άλλοι συνάδελφοί μου ανέπτυξαν υπό αυτές τις συνθήκες. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι στην προσπάθειά σας να ε, επιφέρετε κάποια ε, ηρεμία στους καταθέτες ε, δημιουργήθηκε το αντίθετο φαινόμενο. Οι καταθέτες να καταθέτουν ή να μεταφέρουν τις καταθέσεις τους σε τράπεζες της Κεντρικής Ευρώπης οι οποίες είναι ισχυρότερες και είναι πολύ λογικό να πιστεύουν ότι είναι πιο ασφαλής η κατάθεσή τους σε μια ισχυρότερη τράπεζα. Θα ήθελα λοιπόν να δω πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε κύριε Κρεμαστινέ. Ναι. Το λόγο έχει η κυρία Μπάρμπαρα Λέτσι από την Ιταλική Γερουσία. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Ρεν για την κατάσταση στην Ιταλία. Έχουμε ένα προϋπολογισμό το 40% του οποίου... Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημοσίου χρέους, έχουμε και εμείς πάνω από 10 δις ε, πρωτογενές πλεόνασμα που μειώνει το δημόσιο χρέος. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική σταθερότητα που χαρακτήριζε τη χώρα μας ε, την τελευταία 20 αιτία, διότι υπήρχαν δύο παρατάξεις που εναλλάσσονταν ε, στην εξουσία και που οδήγησαν σε μια εκθετική αύξηση της φορολογικής πίεσης ε, στην Ιταλία, στις επιχειρήσεις και στην οικογένεια και όπου υπάρχει και εχθρότητα από πλευράς των πιστοτικών δομών. Οι τράπεζες ε, προωθούν πολιτικές προς όφελός τους και συνεχίζουν να εφαρμόζουν ε, πολιτικές επιβάρυνσης του δημοσίου χρέους. Μεγάλο κομμάτι του χρέους της Ιταλίας πηγαίνει στις τράπεζες, πηγαίνει στις τράπεζες μας. Πώς λοιπόν αυτή η θεωρητική ανάκαμψη θα προχωρήσει αν όλη αυτή η οικονομική πολιτική διαμορφώνεται βάσει δεδομένων που είναι, όπως έλεγε το πρωί, τελείως ε, θεωρητικά ε, και δεν ελέγχονται από κανένα οικονομικό ε, ιστιτούτο χωρίς να μειώσουμε την φορολογική επιβάρυνση επιχειρήσεων και οικογενειών με αποφασιστικό τρόπο για να προσπαθήσουν να διευρύνουν την παραγωγική βάση που τα τελευταία χρόνια το μόνο που κάνει είναι να, χτυ... να χτυπά τον ε, πολίτη. Δεν έχουμε κυβέρνηση που καταφέρει να διατηρήσει την, που καταφέρει να διατηρήσει την ε, σχέση ελλείμματος με μόνο διαδικασία που είναι εις βάρος των, ε, ε εις βάρος των εργαζομένων και εις βάρος και με κριτήρια τα οποία δεν υφίστανται. Ευχαριστώ. Έχει ο κύριος Πάουλο Μότα Πίντο από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, η Πορτογαλία, όπως προβλέπετε, θα βγει από το πρόγραμμα στις 17 Μαΐου του 2014. Υπάρχει μια συνεχιζόμενη συζήτηση όπου για το κατά πόσο θα χρειαστεί ένα προληπτικό νέο πρόγραμμα μετά την έξοδο ή όχι, για να δεν χρειαστεί. Θα θέλαμε να Μην χρειαστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα εμφανιστεί στο τέλος. Ελπίζουμε ωστόσο ότι η οικονομική εξέλιξη θα καταστήσει περιττό το πρόγραμμα αυτό. Επίσης, υπήρχαν ε, κενά στο σχεδιασμό του προγράμματος μέχρι τώρα. Κάποιοι στόχοι δεν ήταν ρεαλιστικοί, ιδίως του ελλείμματος, που δημιούργησαν σημαντικές κοινωνικές συνέπειες. Η Πορτογαλία, ωστόσο, βγαίνει από το πρόγραμμα και η αξιολόγηση είναι πάντα επιτυχής. Ε, νομίζω ότι εμεί έχουμε καταφέρει να ισορροπήσουμε σωστά την εξηγένση και την ανάπτυξη. Στο μέλλον είναι σημαντικό ωστόσο να ξέρουμε κατά πόσον η ανάπτυξη που έχουμε πετύχει τώρα είναι βιώσιμη λόγω του υψηλού επίπεδου χρέου. Η Τραπεζική Ένωση επίση είναι σημαντική για μα. Θέλουμε να συμφωνηθεί πριν τι ευρωεκλογέ, αλλά ε, με τρόπο που θα επιτρέπει να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τελειώσω με δύο μαθήματα από την κρίση. Πρώτον, να βελτιώσουμε και να διαφυλάξουμε το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαδικασία αυτή. το αίσθημα ότι τα προγράμματα προσαρμογής είναι δική μας δουλειά και η νομιμοποίησή του απαιτούν εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων, περισσότερο από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Στο μέλλον, η προσπάθεια να συζητούμε χρηματο... Ε, τους οικονομικούς στόχους ε, πρέπει να γίνεται νωρίτερα για να μην ε, φαίνεται στην κοινωνία ότι απλώς επιβάλλονται από τα έξω. Επίσης, ο ρόλος της Επιτροπής και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για να επιτρέψουν την ανάπτυξη και να υπάρχει συνένεση και στην ε, πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Η συνένεση υπήρχε στο ξεκίνημα, αλλά σταδιακά διαβρονόταν. Υπάρχει μια πρόταση για συνένεση σε κανόνες δαπανών και ε, ελλείμματος. Στις χώρες όμως όπου γίνονται συζητήσεις, μεγάλες συζητήσεις για γεγονότα και για πολιτικές, όχι δηλαδή αν υπάρχει μια, μια, μια, από, ε, πολιτική αποπληθωριστική και μια ε, έλλειψη της ανάπτυξης, είναι σημαντικό να έχουμε συνεισφορά από τα έξω από την Επιτροπή για να μπορέσει να, η συνένεση αυτή να γίνει σε, μακρο, σε μακρόπνο επίπεδο. Συμβάλλοντας και στην υπέρβαση μελλοντικών κρίσεων. έχει ο κύριος από το Βελγικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, χαίρο που... Εδώ, εδώ είμαι. Χαίρο που μπορώ να συζητώ μαζί σας κύριε Πίτροπε, γιατί συχνά έρχεστε και ζητάτε τις κυβερνήσεις σας, ε, τους λέτε να κάνουμε, μας το εξηγούν αυτό και θα ήθελα να αμφισβητήσω την συνταγή που επιβάλλεται. Βεβαίως χρειάζεται δημοσιονομική αυστηρότητα, λιτότητα. Κανείς δεν μπορεί να ζει εσάι, καμιά χώρα δεν μπορεί να ζει εσάι με χρέη που τα περνάει στο μέλλον, αλλά οι κοινωνικές επιπτώσεις ό,τι αφορά την αύξηση της φτώχειας, την κατανομή του πλούτου, τα μέτρα που επιβάλλονται σήμερα στις συντάξεις, στην ανεργία, στην αγορά εργασία. Ε, μας οδηγούν στο να πιστεύουμε ότι ο προσανατολισμός είναι λάθος και οι στόχοι της Ένωσης εν ώψη του προγράμματος Ευρώπη 2020 για μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους ξεχάστηκαν από τις ε, σύνταγες που επιβάλλουν σήμερα τα κράτη-μέλη μετά από ευρωπαϊκή πίεση και με εντυπωσιάζει πάντα η σκληρότητα των μεταρρυθμίσεων που επιβάλλονται που επιβάλλονται σχεδόν στα κράτη ε, αμφισβητείται η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών που υπάρχει στο Βέλγιο, ενώ αποδυναμώνονται οι μεταρρυθμίσεις ε, που έχουν ξεκινήσει στον τραπεζικό τομέα. Υπάρχουν αδυναμίες στις λύσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ή των ε, φορολογικών παραδείσων που θα, θα μπορούσαν να δώσουν ή μέτρων που θα μπορούσαν να δώσουν νέα έσοδα όπως ο φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Με την ευκαιρία να σας πω ότι αν θέλετε να υπάρχει μια βιώσιμη αποτελεσματικότητα των λύσεων που επιβάλλονται και να αντιμετωπίσουμε την απόρριψη της Ευρώπης από τους συμπολίτε, προσπαθήστε να εξισορροπήσετε την δημοσιονομική πληθαρχία με περισσότερη κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη και μάχη κατά της ε, φοροδιαφυγής. Δεν ξέρω αν αυτό είναι στην ημερήσια διάταξή σας, παρότι ακόμα έχετε λίγους μήνες δουλειάς, δεν ξέρω αν θα ξαναρχίσετε μετά το Μάιο. έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα απαντήσω με τυχαία σειρά. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση του κύριου Ματαπίντο από την Πορτογαλία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα συμπεράσματα που εξάγεται από την εφαρμογή του προγράμματος στην Πορτογαλία μέχρι στιγμής. Συμμερίζομαι τα συμπεράσματά σας, ιδιαίτερα όσον αφορά το αίσθημα οικειοποίησης του προγράμματος. Είδαμε ότι στις χώρες όπου ήταν πιο ισχυρή η οικειοποίηση και όπου η εθνική ενότητα τελικά ε, κυριάρχησε, επέστρεψε η εμπιστοσύνη πιο σύντομα. Και έτσι τέθηκε η βάση για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση. Έχουμε τις περιπτώσεις Ιρλανδίας και Λετωνίας, αλλά και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Επιδεικνύουν ισχυρό αίσθημα οικειοποίησης που βελτιώνει τις πιθανότητες επιτυχίας. Πιστεύω ότι και στην Ελλάδα μπορεί να αυξηθεί το αίσθημα οικειοποίησης, διότι αποτελεί προϋπόθεση για επιτυχία των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Ρωτήσατε, σχετικά με... Ρωτήσατε αν η Πορτογαλία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μια λεγόμενη καθαρή, καθαρή έξοδο ή εάν χρειάζεται κάποια προληπτική ρύθμιση ή είναι ακόμα πολύ νωρίς για να λάβουμε οριστική θέση στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομία, στις χρηματοοικονομικές αγορές, θα αναλύσουμε την κατάσταση κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων και μηνών. Και κάποια στιγμή, μέσα στο χειμώνο ή την άνοιξη, θα καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Πορτογαλίας, με τη ζώνη του ευρώ και τους διεθνείς εταίρους μας. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Κρεμαστινού. Αναφερθήκατε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απομένουν ακόμα να γίνουν πολλά στην Ελλάδα για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα και να μεταρρυθμιστούν οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Πρέπει να προχωρήσουν οι εργασίες και για την υιοθέτηση της νομοθεσίας για το πλαίσιο ανακεφαλοποίησης των τραπεζών ώστε να είναι έτοιμο μετά τις ε, ε, δοκιμές ε, προσωμείωσης ακραίων καταστάσεων των λεγόμενων stress test. Θα πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθούν τα ελληνικά stress test. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα συνεχίζονται και οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο. Στο εγγύς μέλλον, η μεθοδολογία του ενιαίου μηχανισμού παρακολούθησης ε, της ε, Ευρωζώνης θα δημοσιοποιηθεί και μπορεί να ληφθεί υπόψη η ε, μεθοδολογία αυτή κατά την διεξαγωγή των ελληνικών ασκήσεων προσωμείωσης ακραίων καταστάσεων. όσον αφορά τις προσπάθειές σας. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να επαναλάβω τη σημασία του αισθήματο οικειοποίηση. Νομίζω ότι το κόμμα σας συμμετέχει στην ελληνική κυβέρνηση και ένα μάθημα από την κρίση είναι ότι για να πετύχουν οι προσπάθειες μεταρρύθμισης απαιτείται ισχυρό αίσθημα οικειοποίησης ε, της Εθνική κυβέρνηση και του Εθνικού Κοινοβουλίου για να γίνουν οι απαραίτητες ε, μεταρρυθμίσει στην κοινωνία και την οικονομία. Η κυρία Σβέτση αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Ιταλία και τον οικονομικό κατακαιρματισμό. Έχετε δίκιο ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς. Ο χρηματοοικονομικός κατακαιρματισμός αποτελεί εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη και γι' αυτό η Κομισιόν ανέλαβε πρωτοβουλία ήδη πέρσι και πρότεινε ένα σύστημα με το οποίο μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσουμε το κόστος δανεισμού ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δυστυχώς, όπως σημειώθηκε στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, τα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα απαντήσει θετικά σε επαρκή βαθμό. Καλό τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή και να δουν θετικά την εφαρμογή. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης ε, της ε, Τράπεζας ε, της Αγγλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα στοχευμένων μέτρων για, τον, για τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι μπορεί να υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύω ότι πιο γενικά φαίνεται να αποδίδει η προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου που αποτελεί συνδυασμό δημοσιονομικής πολιτικής και πολιτικής ανάπτυξης με κίνητρα. Υπάρχουν και κάποια μη συμβατικά μέτρα. Επίσης αναφέρθηκαν οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης. Αναφερθήκατε και στους φορολογικούς παραδείσους. με τον ε, Διεθνή Συντονισμό Πολιτικής και με τη Μερή ε, συμφωνίας ε, καταφέραμε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια να κλείσουμε παραθυράκια που σχετίζονται με τους φορολογικούς παραδείσους. Στο G20 ασχολούμαστε με αυτό, θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες ώστε να φροντίσουμε να μην έχουμε παραθυράκια, να μην έχουμε φορολογικούς παραδείσου εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερθήκατε στην κοινωνική δικαιοσύνη που θα πρέπει να συνοδεύει την καλή δημοσιονομική πολιτική και ένα πιο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη όπως και οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας μπορεί να ε, οδηγήσει σε, σε καλύτερη σχέση κόστους-όφελους ε, και καλύτερη ε, φροντίδα για τους ασθενείς. Όσον αφορά την οικονομική και νομισματική πολιτική, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Κομισιόν πρόσφατα παρουσίασε μια πολιτική πρωτοβουλία για την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Προσβλέπουμε στην εφαρμογή αυτών σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του φετινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πιστεύω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό περαιτέρω στην ε, επόμενη συνεδρίαση, όπου θα παρευρεθεί και ο κύριος ε, Λάσλο Αντόρ. Πρέπει να γίνει η διάκριση ανάμεσα στα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα βήματα που πρέπει να αναλυφθούν. Για παράδειγμα, μέσοπρόθεσμα, το σχέδιό μας προβλέπει καλύτερο συντονισμό στις αγορές εργασίας ε, της Ευρωζώνης, ενώ μακροπρόθεσμα προβλέπεται η δυνατότητα προϋπολογισμού της Ευρωζώνης ε, που να βοηθάει στην ε, απόσβεση των κλειδονισμών στα κράτη-μέλη. Αυτές, κύριε Πρόεδρε, ήταν οι απαντήσεις μου αυτή τη στιγμή. Νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον τρίτο γύρο. Ελίζα Φερέιρα από το Ευρωκοινοβούλιο. Παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που είστε εδώ για μια ακόμη φορά. Δύο ερωτήσεις έχω να σας απευθύνω. Πρώτη ερώτηση για το χρέος. Αναφέρατε ότι στο τέλος του προγράμματος είχε υπάρξει αύξηση του χρέους κατά 5%, δηλαδή από το 60% στο 90%. Ποια είναι η θέση σας, θα αναλάβει πρωτοβουλία η Κομισιόν με βάση το έργο το οποίο οργανώνεται για την αμοιβεοποίηση ή τέλος πάντων το συντονισμό του τρόπου με τον οποίο ολείται το δημόσιο χρέος ή πιστεύετε ότι αρκεί ε, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, χρυσές μετοχές, τα golden shares. Ζητά από τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τα κράτη-μέλη που είναι σε μνημόνιο να καταργήσουν αυτές τις μετοχές. Οι αρμόδιοι όμως λένε ότι ένα από τα στοιχεία της, ε, των μνημονίων ήταν η ιδιαιτικοποίηση πολύ κρίσιμων τομέων όπως ενέργεια, ε, τηλεπικοινωνίες, ασφάλειες, ε, τράπεζες. Πολλές φορές η πώληση έγινε με πολύ αρνητικούς όρους, σε εταίρους που δεν ήταν και τόσο δημοκρατικοί, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Ποια λοιπόν ήταν αυτά τα κριτήρια για τους στρατηγικούς αυτούς κλάδους, για τις χρυσές λεγόμενες μετοχές και αν αληθεύει ότι η ιδιωτικοποίηση ήταν μεταξύ των όρων που επέβαλε η Τρόικα, διότι λαμβάνουμε τελείως αντιφατικές πληροφορίες. Άλλα μας λέτε εσείς και άλλα μας λένε οι κυβερνήσεις. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Από την Λετωνία ο κύριος Πίμενον Άκπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αναφέρατε τη Λετωνία. Τη χαρακτηρίσατε ένα επιτυχημένο παράδειγμα της ε, δημοσιονομικής πολιτικής. Ε, το μυστικό όμω της επιτυχίας της Λετωνίας ε, είναι πάρα πολύ απλό. Η δραστηριότητα της λετωνικής οικονομίας ήταν ανάλογη της ύφεσης μετά την μεγάλη ύφεση στις ΙΠΑ και την κρίση της Αργεντινής ήταν η τρίτη φορά που είχαμε μια τέτοια ύφεση. Πρέπει να σας πω ότι ναι μεν έχουμε κάποια θετικά στοιχεία στις μακροοικονομικές εκθέσεις για τις επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι το χρέος οφείλονταν στην προκυκλική πολιτική που εμπνεύστηκε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν και την στήριξε και η λετωνική κυβέρνηση που ήθελε να οδηγήσει με κάθε τίμημα την Λετωνία στην Ευρωζώνη. Και υπήρξε εσωτερική υποτίμηση. Μειώθηκαν οι μισθοί, χάθηκαν θέσεις εργασίας, μειώθηκαν οι ε, δημόσιες δαπάνες για να πετύχουμε το στόχο αυτό. 25% λοιπόν μειώθηκε το ΑΕΠ, τεράστιο χρέος, μείωση της απασχόλησης κατά 20%. Μιλάμε τώρα για όλο και περισσότερους ε, μακροπρόθεσμα ανέργους. Αυτό είναι λοιπόν ε, το... η επιτυχία της Λετωνίας. Πρόεδρος, πρέπει να σας ε, ενημερώσω ότι οι παρουσιάσεις όλων των ομιλητών που λαμβάνουμε θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της συνέλευσής μας στο www.europarl.europa.eu είπε 2014. Στην ιστοσελίδα της συνέλευσης θα αναρτώνται, επαναλαμβάνω, όλες οι ομιλίες που λαμβάνουμε τουλάχιστον. Επίσης, έχω, ε, εδώ θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Και επειδή είναι πολλοί οι ομιλητέ, θα περιοριστούν όλοι στα δύο λεπτά. Θα είμαι αυστηρό. Ο κύριο Καρέας από τη Γαλλία έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Και εντάχει. Δεν θα ενδώσω στην εύκολη λύση της κατηγορίας της Επιτροπής ούτε στο να δείχνω με το δάχτυλο την Επιτροπή ως υπεύθυνη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας. Διότι η προσανατολισμοί της επιτροπή επικροτούνται και υλοποιούνται και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα η ευθύνη εν τέλει είναι ευθύνη πολιτική που ασκείται κυρίως μέσω των συστάσεων, επί των συστάσεων. Επίσης διότι υπάρχει και ευθύνη των κυβερνήσεων στην κρίση, πρέπει να το πούμε αυτό, με ευθύνη γιατί κάποιοι επέτρεψαν να ξεφύγει με τελείως ανεύθυνο τρόπο το έλλειμμα. Μην κατηγορούμε λοιπόν την Επιτροπή υπερβολικά, παρότι είναι αλήθεια και αναφέρθηκε ήδη ο τρόπος με τον οποίο περιγράψατε την δράση των Επιτροπών τα τελευταία χρόνια, κύριε Ρεν, ε, δείχνει ότι και εσείς αναθεωρήσετε κάποια πράγματα σε σχέση ιδίω με τον ρυθμό προσαρμογή. Η ερώτηση που θέλω να σας θέσω, κύριε Ρεν, είναι απλή. Πώς τη στιγμή που ξεκινά η ανάκαψη, αλλά είναι εξαιρετικά ευάλωτοι και υπάρχουν πολύ σημαντικές αβεβαιότητες, πώς θα συνοδεύουμε την ανάκαψη αυτή σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαθροτικών αλλαγών. Αναγκαίες μένα, αλλά έχουν και κόστος σε κάποιες χώρες. Πώς συνοδεύουμε την ανάκαψη αυτή, μήπως χρειάζονται και άλλα νέα εργαλεία, ιδίως σε επίπεδο ε, προπολογισμού είτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είτε τη Ευρωζώνη για να αντιμετωπιστούν αυτέ οι ασυμμετρικέ επιλογέ και να μπορέσει να παγιωθεί η ανάκαμψη. Τι άποψη έχετε περί αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καβερέιτα από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Ρεν, ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ μαζί μας. Δεν συμφωνώ με την λαμπερή εικόνα που έχετε για τις ε, πολιτικές ε, εξυγένσεις και τις πολιτικές της Τρόικας. Αν δείτε το σχέδιο έκθεσης της, ε, του Ευρωπαϊκού Βιβλίου, η Πορτογαλία το 2007, την τελευταία χρονιά δηλαδή πριν τη χρηματοοικονομική κρίση, είχε 62% έλλειμμα, ε, χρέος, 3% έλλειμμα ενώ η οικονομία αναπτυσσόταν με ρυθμό άνω του 2%. Λόγω της έλλειψης επίκαιρης και έγκαιρης ανταπόκρισης της Ευρώπης στην κρίση και λόγω της πολιτικής αστάθειας η Πορτογαλία υποχρεώθηκε σε μια πολιτική προσαρμογής. Η συμφωνία αυτή εφαρμόστηκε με σκληρότερα μέτρα από ό,τι προβλεπόταν στο αρχικό μνημόνιο. Οι πολιτικές λιτότητας υπερδιπλασίασαν τις προβλέψεις. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η Τρόικα ως τεχνικό εργαλείο αρνήθηκαν να συζητήσουν χρήσιμα με τους κοινωνικούς εταίρους της Πορτογαλίας και το κοινοβούλιο της χώρας. Τώρα, μπορείτε να μιλάτε για τα δημοσιονομικά, για τα νομισματικά ζητήματα. Δείτε όμως την πραγματική οικονομία, την, ε, τον κοινωνικό τομέα. Πραγματικά η οικονομία της Πορτογαλίας είναι τώρα χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από 2,5 χρόνια. Και υπάρχει ευρεία κοινωνική συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών, εργαζομένων κατά του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε το πρόγραμμα προσαρμογής. Έχουμε τρία χρόνια ύφεση, την χειρότερη ανεργία σε εποχές δημοκρατίας. Η Πορτογαλία είναι μια ισχυρά, εμφαντικά φιλοευρωπαϊκή χώρα. Εμείς ξεκινήσαμε με οικονομική κρίση, έχουμε, βιώνουμε τώρα κοινωνική κρίση και δεν περιμένουμε μετά τις ευρωεκλογέ να έχουμε πραγματική εμπιστοσύνη στην Ευρώπη λόγω των πολιτικών της Ένωσης. Θέλουμε μια Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη, χωρίς, όχι όμως μια Ευρώπη χωρίς συζητήσεις με τους πολίτες, όπου οι πολίτες κλειδώνονται έξω από τις συζητήσεις, όπως συνέβη πριν από 2,5, αυτά τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Συνέβησα από την Γερμανία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. αν δεν κάνω λάθος, το θέμα σήμερα είναι σκέψεις για καλύτερη υποπτία του προϋπολογισμού των δημοσιονομικών ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι καλύτερο είναι να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό και να θέτουμε ερωτήσεις προς τον κύριο Ρεν που αφορούν την βελτίωση της ε, δημοσιονομικής εποπτείας. Ε, νομοθετικά μέτρα όπως είναι η δέσμη των 6 ε, μέτρων, ε, των 2 μέτρων, το ΣΥΞΠΑΚ και το ΤΟΥΠΑΚ δηλαδή και άλλα. Στα χρόνια μετά την εισαγωγή του ευρώ είδαμε ότι η εποπτεία δεν λειτουργήσε αρκετά καλά. Τώρα έχουμε το δημοσιονομικό σύμφωνο και πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εφαρμοστεί το σύμφωνο αυτό και μαζί με την Κομισιόν ε, να ε, εποπτεύουμε την εφαρμογή. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει πώς μπορεί να βελτιωθεί η εποπτεία αυτή. Ο κύριος Ρεν παρουσίασε την ε, ανάπτυξη ως έχει, είναι θετική. Έχουμε μείωση των χρεών, ε, δημοσιονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Αυτά τα βρίσκω καλά και σωστά, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει τους στόχους του Μάστριχτ. Ε, στο Μάστριχτ προβλέπεται έλλειμμα το πολύ 3% δεν έχουμε πετύχει καθόλου τους στόχους αυτούς ακόμα, γι' αυτό θα πρέπει να γίνει καλύτερη η εποπτεία, η δημοσιονομική εποπτεία. Από γερμανικής πλευράς ε, θεωρούμε ότι η δημοσιονομική εξυγίαση δεν είναι το αντίθετο της ανάπτυξης του αντίον. Ε, είναι ο καλύτερος τρόπος ε, να κινητοποιηθεί η ανάπτυξη. Οι νέες θέσεις εργασία δημιουργούνται εκεί όπου οι επενδυτές έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον της χώρας. Αποτελεί λοιπόν ε, απαραίτητη προϋπόθεση για την ε, οικονομική ανάπτυξη. Μία τελευταία παρατήρηση. Η καλύτερη υποπτία είναι απαραίτητη. Όταν ακούω τις παρεμβάσεις των Ελλήνων ε, συναδέρφων ε, που είναι κατά αυτόν που λέει ο κύριος Ρέν, ποιον πρέπει να πιστέψω εγώ, τον κύριο Ρέν ή τους Έλληνες συναδέρφους, ε, διότι αν δεν λειτουργεί η εποπτεία σας όπως λένε οι Έλληνες συνάδελφοι, εάν δεν λειτουργούν τα προγράμματα, αναρωτιέμαι εάν η Κομισιόν στόχο έχει να προτείνει σε όλους μας τη συνέχιση του προγράμματος που αφορά την Ελλάδα. Ποιον πρέπει να πιστέψω τελικά. Ευχαριστούμε. Ε, ο κύριος, το λόγο έχει ο κύριος ε, Ζωάο Καλάμπρα από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις για τον κύριο Ρεν. Πρώτον, κάνετε δηλώσεις, συνεχίζετε να κάνετε δηλώσεις που δεν ανταποκρίνονται στα γεγονότα. Για την δημοσιονομική κρίση στην Πορτογαλία, για παράδειγμα. Θα ήθελα να πω το εξή. Πώ μπορεί η Επιτροπή να λέει ότι υπερδαπάνισε η Πορτογαλία ενώ το 2008 και έχω μπροστά εδώ το σχετικό έγγραφο τον Ιούνιο του 2008 μετά από σύσταση τη επιτροπή, στο Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έλλειμμα τη Πορτογαλία ήταν κάτω από το 3% του ΑΕΠ με βιώσιμο και αξιόπιστο τρόπο. Εγκαταλείψαμε την, το 2008 την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Με δεδομένα αυτά, πώ μπορείτε να λέτε ότι η κρίση στην Πορτογαλία ήταν κρίση αύξηση των δαπανών. Επίσης, στις τριμενιαίες εκθέσεις Επιτροπής, αν δείτε τις, ε, τα στοιχεία για την εσωτερική ζήτηση, η Πορτογαλία μετά τη Γερμανία ήταν η χώρα στην Ένωση όπου η δημόσια κατανάλωση δεν αυξανόταν, παρότι υπήρχε ανάπτυξη. Με αυτά τα δεδομένα μπορείτε να μας εξηγήσετε λοιπόν σε ποια στοιχεία στηρίζεται τις θέσεις σας ότι η Πορτογαλία είχε μια δημοσιονομική κρίση πριν τη γενική χρηματοοικονομική κρίση. Ο στόχος της ε, Πορτογαλίας πρέπει να είναι η ανάπτυξη. Ε, το βασικό της πρόβλημα ήταν η ανάπτυξη. Είχε αναπτυχθεί σχετικά χαμηλά την τελευταία δεκαετία. Μια φτωχή χώρα που πρέπει να επενδύσει σε εκπαίδευση, σε έρευνα, πώς μπορεί να κρατήσει ε, ανάπτυξη σαν ποσοστό του ΑΕΠ όταν περικόπτουμε τις δημόσιες επενδύσεις, την ανανεώσιμη ενέργεια, την εκπαίδευση, την έρευνα και ανάπτυξη. Περιέργω, σύμφωνα με στοιχεία από την Επιτροπή σας, από το, τη Γενική σας Διεύθυνση μάλιστα, η, το ΑΕΠ τη Πορτογαλίας κατά τη διάρκεια του προγράμματο μειώθηκε. Με αυτά τα δεδομένα θα ήθελα να ρωτήσω πώ δικαιολογείται μια σειρά δηλώσεων που συνεχίζει να κάνετε για τη χώρα μου. Ευχαριστώ. Είναι ο κύριος Φραντζέσκο από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χτες ολοκληρώθηκαν οι υποψηφιότητες για το λεγόμενο Fiscal Council, το Διοικητικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στη χώρα μου ε, καθυστέρησαν να ορίσουν τα μέλη που τις αντιστοιχούν. Εν ώψη της προετοιμασίας του κανονισμού, το κίνημα των πέντε αστέρων που εκπροσωπώ εδώ, έδωσε έμφαση σε μια σειρά θεμάτων. Διαφάνεια των βιογραφικών, ανεξαρτησία του οργάνου και υποχρέωση των, ε, υποχρέωση των υποψηφίων να παρουσιάσουν το ποινικό μητρό τους. Μόνο το τελευταίο έγινε δεκτό από το Κοινοβούλιο και θα ήθελα να θέσω την εξή ερώτηση στον Επίτροπο κύριο Ρεν. Πώς βλέπει τον ρόλο του οργάνου αυτού και από τεχνικής απόψεως και από πολιτικής απόψεως. Ποια στοιχεία πρέπει να παράσχει, σε ποιες παραμέτρους θα εδράζει η ευθύνη του οργάνου αυτού για να δημιουργηθεί ένα στάνταρ και να αποφασίσει κατά πόσο πραγματικά η Ένωση προχωρά προς μια ανάκτηση από την ύφεση ή αν κάθε φορά θα πρέπει να αφήνουμε την ερμηνεία αυτή στους διάφορους ε, επιτρόπους που μας επισκέπτονται. Και τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε ότι τις χώρες που έχουν ήδη ενσωματώσει τώρα όργανο αυτό θεσμικά. Κάποιες χώρες που είναι πιο μπροστά από την Ιταλία στη δημιουργία αυτού του Fiscal Council. Τι θεωρούν ότι μπορεί να βελτιωθεί στη χώρα για να είναι καλύτερος αυτός ο θεσμός. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Λέντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα πολύ εύστοχα ερωτήματα. Θα ξεκινήσω από το τέλος, ε, γιατί θυμάμαι πιο καλά τα τελευταία ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Κοριέλου και το ερώτημά του για την ε, φύση των ανεξάρτητων δημοσιονομικών συμβουλίων. Ε, είναι πολύ σημαντικό ερώτημα πράγματι και αυτό αποτελεί και ένα ουσιώδη στοιχείο για την αποτελεσματική δημοσιονομική επιτήρηση, ώστε να έχουμε μεσοπρόθεσμα βιώσιμα οικονομικά. Και εντάσσεται το στοιχείο αυτό Δεν μ' αρέσει βέβαια αυτή η ορολογία, αλλά σε αυτό το εξαπλό πακέτο, ε, το six-pack, ε, και στο δημοσιονομικό σύμφωνο, το Fiscal Compact, που συμφωνήθηκαν από τα κράτη-μέλη. Μου κάνατε μια έτσι πολύ ευθεία ερώτηση. Τι είδους δημοσιονομικών συμβουλίων συνιστώνται στο πλαίσιο αυτό. Θα σας απαντήσω. Υπάρχουν παραδείγματα που συνάδουν με τις συνθήκες και με τις διδάξεις του Δημοσιονομικού Συμφώνου και μπορούμε να τα αναφέρουμε, αξίζει τον κόπο. Αν εγώ ήμουν βουλευτής οποιοδήποτε κράτους μέλους, ε, θα έβαζα ως παράδειγμα την Ολλανδία ε, και το γραφείο του Γιάνν Τίμπεργεν, που ήταν ε, βραβευμένος το 69 με βραβείο Νομπέλ, ο πρώτος που πήρε. Βέβαια αυτό το συμβούλιο νομίζω συστάθηκε τη δεκαετία του 50, αν δεν με μου, και έχει την ευθύνη του να κάνει ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις και δημοσιονομικές εκτιμήσεις. Το σύστημα στην Ολλανδία πηγαίνει σε τόσο μακριά ώστε και τα οικονομικά προγράμματα ε, των ε, κομμάτων πριν ε, κατέχουν σε εκλογές αναλύονται από αυτό το όργανο, το CPB. Τι είναι λοιπόν ουσιώδες. Με τον ένα τον άλλο τρόπο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα αυτά τα συμβούλια και να προβαίνουν σε ανεξάρτητες μακροοικονομικές ε, προβλέψεις. Κατά το παρελθόν αντιμετώπισαμε τεράστια προβλήματα στον τομέα αυτό και γι' αυτό δεν υπήρχε ουσιαστικά αποτελεσματική εποπτεία, αποτελεσματική επιτήρηση. Μέχρι που ξέσπασε η κρίση. Ακόμη και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες δεν μπορούσαν να ανοιχτευτούν. Πρέπει λοιπόν να είναι ανεξάρτητα τα δημοσιονομικά συμβούλια για το στόχο αυτό. Και επίσης είναι πολύ καλό που κάνουν και αξιολογήσεις των διαφόρων μέτρων. Πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστα και πιστικά. Σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική επιτήρηση, το ρωτήμα Μπάθρας, Επαναλαμβάνω αυτό που είπα για τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβουλία. Συμφωνώ πάντω μαζί σα. Και έχω και εγώ την εντύπωση ότι πιο πολύ αφορούσε την οικονομική κατάσταση των χωρών που είναι σε πρόγραμμα προσαρμογή. Δεν αφορά τόσο τη μεθοδολογία δηλαδή τη δημοσιονομική εποπτεία. Γνωρίζω, γιατί υπήρξα, διατέλεσα μέλο και Εθνικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γνωρίζω ότι στα κοινοβούλια και ιδίω ε, στι δημόσιε συνεδριάσει μπορεί κανείς ε, να ρωτήσει και να σχολιάσει επί παντός επιστητού. Εγώ προσπαθώ να απαντήσω ε, όσο με επιτρέπουν οι γνώσεις μου. Νομίζω όμως ότι είναι καλό πράγματι να εστιάσουμε σε αυτή τη συνεδρία στην δημοσιονομική αποπτία. Και επειδή με ρωτήσατε, γιατί μιλάμε για τις δημοσιονομικές πολιτικές εδώ, η έμφαση πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση, στην εφαρμογή των ενισχυμένων αυτών πλαισίων οικονομικών και ε, προγραμμάτων και δημοσιονομικής εποπτείας που καταρτήσαμε τα τελευταία χρόνια. Και το επόμενο κοινοβούλιο, η επόμενη κομισιόν θα πρέπει να τα αναθεωρήσει όλα αυτά. Γιατί στόχος είναι η απλούστευση. Και να είναι πιο κατανοητά όλα αυτά από την κοινή γνώμη. Αλλά και από τους ευρωβουλευτές και από τα μέλη της ε, κομισιόν. Πολύ σωστά λέτε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για επενδύσεις, για θέσεις εργασίας είναι η εμπιστοσύνη. Καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία και στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Και αυτό κυρίως χάρη σε τρεις παράγοντες από το 2012, όταν τέθησαν τα θεμέλια για την οικονομική ανάκαμψη. Πρώτος παράγοντας, η βελτιωμένη αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών μελών όπως καταδεικνύεται από το γεγονός ότι μειώθηκαν τα δημοσιονομικά ελλείμματα από το 7% στο 3%. Δεύτερον, αποφασιστική δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη σταθεροποίηση ε, των χρηματαγορών και των αγορών ομολόγων μετά το 2010. Και τρίτον, ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση που έχουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη. Αυτό παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για την συνεχή εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών μεσοπρόθεσμα, αλλά και για την επιτυχημένη πρόθεση των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Αυτοί οι τρεις παράγοντες άλλαξαν το σκηνικό στην ε, διαδικασία λήψεως αποφάσεων, άλλαξαν το κλίμα, τη διάθεση στην Ευρώπη από το 2010 και μετά. και παρότι υπήρξαν πολιτικές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, δεν συντάραξαν ε, τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Καλάμπα ανέφερε την πορτογαλική περίπτωση. Ακούσαμε αρκετά σχόλια για την Πορτογαλία στις παρεμβάσεις. Αναφερθήκατε στην φύση της κρίσης. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας είπατε ότι η κρίση ήταν συνδυασμός ε, επιβραδυμένης ε, ανάπτυξης και υπερβολικού ιδιωτικού και δημοσίου χρέους. Κάτι που έκανε την Πορτογαλία να ζητήσει οικονομική ενίσχυση τελικά. Η κυρία Φερέιρα και άλλοι αναφέρθηκαν στην οικονομική κατάσταση. Η αύξηση της ανεργίας είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής της πορτογαλικής οικονομίας. και κάποια μετατόπιση, μετακίνηση του εργατικού δυναμικού. Υπήρχαν βέβαια και εξωγενείς παράγοντες, εξωτερική ζήτηση, η συμπεριφορά των χρηματαγορών. Ελήψη όμως προγράμματος θα ήταν πάρα πολύ χειρότερες οι κοινωνικές επιπτώσεις. Και σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες πιέσεις και που δεν έχουν ένα ανεπτυγμένο πρόγραμμα παροχής βοήθειας, Βλέπουμε αντίστοιχες ε, καταστάσεις. Σίγουρα η ανεργία είναι πρόβλημα και είναι και ένας από τους βασικότερους στόχους ε, των προγραμμάτων. Και είναι και στόχος των περισσότερων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες μάλιστα έχουν ε, εγκριθεί και από τους κοινωνικούς εταίρους. Ο κ. Καμπρίτα κάποια στιγμή μίλησε για την επιδείνωση της κρίσης στην Πορτογαλία λόγω της καθυστερημένης ευρωπαϊκής αντίδρασης. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ήταν καθυστερημένη και η εθνική αντίδραση. Διότι ναι μεν ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2011 το μνημόνιο στην Πορτογαλία. Θυμάμαι όμως τις πρώτες συζητήσεις που είχαμε τον Υπουργό Οικονομικών της Πορτογαλίας τον Ιούνιο του 2010, ένα χρόνο δηλαδή νωρίτερα, για ένα ενδεχόμενο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, διότι βλέπαμε ότι η οικονομική κατάσταση της Πορτογαλίας αποδυναμωνόταν. Κατά την άποψή μου, όσο πιο γρήγορα αντιδρούσε η Πορτογαλία, τόσο καλύτερα θα τα καταφέρνε να επανεξορροπούσε την κατάσταση χωρίς ένα επώδυνο πρόγραμμα προσαρμογής. Και θα ήταν καλύτερα να το κάνει πριν βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο τον Απρίλιο 2011. Η κυρία Φερέιρα μίλησε για την αμοιβεοποίηση του δημόσιου χρέους. Επ' αυτού ξέρετε ότι έχει συγκροτηθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, και με το Συμβούλιο και θα παρέχει υποστήριξη σε ό,τι αφορά το Ταμείο εξαγορά του Δημοσίου Χρέου. Πριν τα τέλη Μαρτίου, αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι σε εξέλιξη σχετικέ εργασίε. Ο Πίμενον από τη Λετωνία είπε σωστά ότι συνεργαστήκαμε με την ε, λετωνική κυβέρνηση. Και έχετε δίκιο ότι επέλεξε η Λετωνία το δρόμο της εσωτερικής υποτίμησης αντί της εξωτερικής υποτίμησης. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που έχει μακρά ιστορία εξωτερικών υποτιμήσεων και πρέπει να σας πω ότι αν δεν είναι σε κρίση οι χρηματοπιστωτικές αγορές, ίσως αυτό να είναι πιο εύκολο. Αλλά με την ολοκλήρωση των αγορών αυτό καθίσταται όλο και πιο δύσκολο και όλο και πιο επώδυνο σε σχέση με το παρελθόν. Δεν ε, πρόκειται για περίπατο σε καμία περίπτωση μια τέτοια επιλογή. Αυτός ε, ήταν ο σωστός τρόπος, η Λετωνία τα κατάφερε. Κατάφερε να αναστρέψει τα πράγματα και τα τελευταία χρόνια να έχει γυρίσει την κατάσταση. Επίσης ο μίλησε για την ευθύνη των κυβερνήσεων και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Πράγματι είναι ευθύνη των κρατών μελών και των κυβερνήσεών τους, των κοινοβουλίων τους, ε, το να εξασφαλίσουν ότι οι οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών βρίσκονται σε βιώσιμο μονοπάτι. Είναι εύθραυστη ακόμη ανάκαμψη, γι' αυτό θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων για να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την απασχόληση. Θα πρέπει να επιδιορθώσουμε ε, τα οικονομικά, να καταπολεμήσουμε τον ε, κατακαιρματισμό των αγορών, να ε, υλοποιήσουμε στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας των νέων, ένα πρόβλημα που πλήττει πολλά κράτη-μέλη. Και όλα αυτά σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση στην Ευρώπη, οι ισχυρέ οικονομίε, η Γερμανία πρέπει να ενισχύσει την εσωτερική, την εγχώρια ζήτηση και να προωθήσει τι δημόσιε επενδύσει. Η Γαλλία, απ' την άλλη, ε, θα πρέπει να προωθήσει τι οικονομικέ μεταρρυθμίσει ε, για την ανταγωνιστικότητα, για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το ίδιο βέβαια και για την Ιταλία, αλλά και για άλλε χώρε. Αυτό είναι ένα συμπληρωματικό συνδυασμό μέτρων με τα οποία θα έχουμε καλύτερη στήριξη για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη και αυτή τη σύσταση έχουμε διατυπώσει στα εν λόγω κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν απάντησε στην ερώτησή μου ο Επίτροπος για τα golden share και την ιδιωτικοποίηση σε χώρες που βρίσκονται μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση. αν θεωρεί ο πρόεδρος ότι αυτό είναι κομμάτι των συζητήσεων παρακολουθής της ε, δημοσιονομικής πολιτικής, ναι. Εάν ε, μπορεί να καλυφθεί ή να απαντηθεί. Ήδη απάντησα στο Στρασβούργο στην ακρόαση για το ίδιο θέμα. Εκτός μικροφώνου. Να σας απαντήσω τότε. Η ευθύνη απόφασης για το μνημόνιο συνεννόησης ανήκει στα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο κάθε χώρας σε διαβούλευση με τους εταίρους και τα τρία θεσμικά όργανα ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Εθνικό Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απόφαση των κυβερνήσεων, ε, η απόφαση ανήκει στις κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για τις αποφάσεις αυτές. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Ρεν, ευχαριστώ που θα κάτσετε και για την επόμενη συνεδρίαση μαζί μου για την υλοποίηση του, Ευρω... του κύκλου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2013 για τις προτεραιότητες για το τρέχον έτος του 2014. Θέλω να καλωσορίσω εξ ονόματος ε, ως συμ Πρόεδρο τον κύριο Αλέξανδρο Δερμετζόπουλο, μαζί με τον, κύριο, με τον συμπρόεδρο κύριο Αλέξανδρο Δερμετζόπουλο, τον επίτροπο κύριο Λάζλο άντρο που έρχεται, τον Φίλιπ Ντεμπέκερ που θα μιλήσει αμέσω μετά ω εισηγητή τη οικονομική επιτροπή, για την ετήσια έκθεση ανάπτυξη και την Γκουτιέρε Πιτέτο ω εκπρόσωπο τη επιτροπή απασχόληση για το της ε, εγγύησης ε, για το AGS, για την εγγύηση νέων, όπου μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις, αλλά για να το κάνετε αυτό πρέπει να συμπληρώσετε τα έντυπα ομιλίες που έχετε μπροστά στο τραπέζι σας. Κύριε Επίτροπε, θα ξεκινήσουμε με εσάς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκπόνηση της ημέρησιας διάταξης της συνέδριαση. αυτής. Βέβαια, θα πρέπει να με αντέξετε περισσότερο. Θα προσπαθήσω να αποφύγω να επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν ε, στην, ε, στο προηγούμενο κομμάτι αυτής της ε, διάσκεψης και θα επικεντρωθώ στην μελέτη για την ανάπτυξη το 2014 που καλύπτει ε, όπως καταλαβαίνετε, τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα. Θα ήθελα καταρχάς όμως να θέσω το πλαίσιο της ε, οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη, το οικονομικό πλαίσιο της Ευρώπης. Και θα το κάνω αυτό λέγοντας ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου έτους, ε, το οποίο μας έχει παρουσιάσει ενθαρρυντικά σημάδια ανάπτυξης στην Ευρώπη. Είδαμε ότι κάποιοι δείκτες έχουν επανέλθει στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο και οι προβλέψεις μας λένε ότι θα υπάρξει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ε, παραμένουν όμως κάποιες ε, σημαντικές ε, προκλήσεις, ιδιαίτερα ως συνέπεια των αβάσταχτα ψηλών επιπέδων ανεργίας σε κάποια κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν απαραίτητη η συνέχιση των προσπαθειών. Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2014 είναι το θέμα της συζήτησης σήμερα. Η διαδικασία αυτή έχει περάσει τώρα στον τέταρτο κύκλο και συνεχίζει να παραμένει το βασικό κομμάτι της ε, αναζήτησης της Ευρώπης ε, ανάπτυξης και ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Να σας παρουσιάσω τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο το 2014. Καταρχάς, θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την εξυγίανση της δημοσιονομικής κατάστασης. Η ε, εμπιστοσύνη επιστρέφει, τα ελλείμματα έχουν μειωθεί στο μισό. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, ποιότητα των μέτρων, ιδιαίτερα της φορολογίας, όχι αυξάνοντας ε, τους φόρους, αλλά με φορολογικές μεταρρυθμίσεις ε, που θα βελτιώνουν τα κίνητρα και τις ε, προοπτικές ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και ε, βιώσιμες δαπάνες στην κοινωνική ασφάλιση, την καινοτομία και την υποδομή. Η μελέτη αυτή παρουσιάστηκε πριν κάποιες εβδομάδες, στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς και διατηρεί την ίδια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως και πριν. Ταυτόχρονα τονίζονται οι νέες προκλήσεις που εμφανίζονται τώρα κατά τη φάση της ανάκαμψης. Είναι σημαντικό να αποκατασταθεί ο δανεισμός από τις τράπεζες στην πραγματική οικονομία. Ο κατακαιρματισμός όμως εμποδίζει ακόμα τις εταιρείε να λάβουν τους απαραίτητους πόρους. Έχουμε κάνει πολλά στην Ευρώπη, δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως όμως ακόμα η εμπιστοσύνη και σε αντίθεση με τα πρώτα χρόνια της κρίσης, η αβεβαιότητα στους ισολογισμούς σήμερα δεν έχουν τόσο πολύ να κάνουν με τοξικά περιουσιακά στοιχεία όπως ε, ίσχυε πριν 4-5 χρόνια. Η αβεβαιότητα συνδέεται με τη ε, διαδικασία οικονομικής προσαρμογής, δημοσιονομικής προσαρμογής. Γίνονται ασκήσεις προσωμείωσης ακραίων καταστάσεων, stress test και η Τραπεζική Ένωση θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο του θεματολογίου μεταρρύθμισής μας. Βραχυπρόθεσμα θα είναι και πάρα πολύ σημαντικό να μειωθούν ε, να μειωθεί το χρέος των νοικοκυριών ε, και θα πρέπει επίσης να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. Χρειάζεται λοιπόν παραγωγικές επενδύσεις ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στην βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στις επικείμενες προτάσεις του κυρίου Μπαρνιέ και δικέ μου που έχουν να κάνουν με τι μακροπρόθεσμε επενδύσει στην Ευρώπη. Ε, η πρόταση αυτή βασίζεται ε, σε ευρία διαβούλευση με ομάδες ενδιαφορεμένων στην Ευρώπη. Θα πρέπει επίσης να στηρίξουμε τις δυνατότητές μας για καινοτομία. Θα πρέπει να φροντίσουμε το εργατικό δυναμικό μας να έχει τις απαραίτητες δεξιότητες. Αυτό είναι απαραίτητο για να καταπολεμηθεί η ανεργία και οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης. Ο συνάδελφος και φίλος Ελλάς Λοαντόρ θα αναφερθεί στο θέμα αυτό, το οποίο βρίσκεται πολύ ψηλά στο θεματολόγιο μας. Η ανεργία έχει σταθεροποιηθεί, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλή η ανεργία των νέων, καθώς και η ανεργία διαρκείας. Και αυτό απαιτεί άμεση προσοχή από την πλευρά μας. Θέλουμε να επικεντρωθούμε στην κοινωνική δικαιοσύνη που θα πρέπει να συνοδεύει ε, ε, τα σταθερά δημοσιονομικά και θα πρέπει να προλάβουμε την ε, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και έτσι να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα και περισσότερη δικαιοσύνη. Επίσης, θα πρέπει να συνεχίσουμε τον εξυγχρονισμό των δημοσίων διοικήσεων. Έχουν ε, αναλυφθεί πρωτοβουλίε για να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση. Σε πολλά μέρη μεταφερόμαστε σε επιγραμμικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες της Κομισιόν είναι να συνεργαστούν με τις διοικήσεις των κρατών μελών ε, για να έχουμε αποτελέσματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, αξιότιμοι βουλευτές, ε, σημαντικό μέρο του θεματολογίου μα για να περάσει η Ευρώπη από μια εύθραυστη ανάκαμψη σε βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να επιλύσουμε τις ε, δημοσιονομικές ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η διαδικασία αυτή λοιπόν δικαίως παίζει κεντρικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και αξίζει την προσοχή μας. Είμαι βέβαιος ότι και στις εθνικές διαδικασίες, στα Εθνικά Κοινοβούλια των Κρατών Μελών θα ληφθεί αυτό επαρκώς υπόψη. Ο μηχανισμός, ε, η έκθεση του μηχανισμού κατανομής φέτος ε, ε, δημοσιεύθηκε μαζί με την ετήσια έκθεση ανάπτυξης. Σε 16 κράτη επελέγησαν για να αναλυθεί περαιτέρω η κατάστασή τους και ετοιμάζουμε μια εις ανάλυση των 16 χωρών αυτών. Πράγμα απαραίτητο για να αποφασιστεί εάν υπάρχουν ε, ή όχι ανισορροπίες και τι είδους πολιτικές χρειάζονται για να αποκατασταθεί η ισορροπία. Η έκθεση μας δείχνει ότι αρκετά κρατημέλη σημειώνουν πρόοδο στην ε, μείωση του ελλείμματος και χώρες όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία ωστόσο απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες από τις πλεονασματικές χώρες για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες αποκατάστασης της ισορροπίας στην, στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό δεν έχει απλά να κάνει με τη μείωση δαπανών ε, και με τα χρέη. Θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν τα μονίμως υψηλά πλεονάσματα οφείλονται σε ελλείψεις της πολιτικής ε, ή της αγοράς. Στην ουσία, ο στόχος μας είναι η Ευρωζώνη στο σύνολό της ε, να γίνει πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και να είναι έτσι περισσότερο ικανή να παράγει βιώσιμη ανάπτυξη και υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης στην Ευρώπη. Μπορώ να σας ενημερώσω ότι η Κομισιόν θα δημοσιεύσει αυτή την εισβάθος ανάλυση κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης, το πιθανότερο τον Μάρτιο φέτος. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, να κλείσω λέγοντας ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2014 προχωρά. Πολλά έχουν γίνει στην Ευρώπη για τη μεταρρύθμιση των οικονομιών μας, των κοινωνιών μας, των δημοσίων διοικήσεών μας. Βλέπουμε οικονομική ανάπτυξη, αλλά απαιτούνται ακόμα πολιτικές δράσεις η επιτυχία του Ευρωπαϊκού εξαμίου, η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Εξαμίνου θα βοηθήσει την Ευρώπη να περάσει στην βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι κάτι που απαιτεί τη δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων ομάδων και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν και πρέπει κατά τη γνώμη μου να παίξουν σημαντικό ρόλο, ζωτικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Προσβλέπω λοιπόν στη σημερινή συζήτηση πάνω στην ε, ετήσια έκθεση ανάπτυξης για το 2014. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 10 λεπτά ο κύριος Λάζλο Άντορ. Κυρίες και κύριοι αξιότιμοι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το τέταρτο ευρωπαϊκό εξάμεινο πραγματοποιείται σε μια εποχή που η οικονομική οικονομία παρουσιάζει πράγματι σημάδια ανάκαμψη. Όπως όμως προείπε και εξήγησε ο επίτροπο Όλη Ρέν, είναι μετριοπαθή και καθόλου ομοιόμορφη σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η ανάκαμψη. Η ανεργία έχει σταθεροποιηθεί στο 26 ε, δεν βλέπουμε να υπάρχει όμως τάση σταθερή για αύξηση ε, της απασχόλησης. Ε, τα τελευταία χρόνια δεν πετύχαμε πολλά στον τομέα της απασχόλησης. Η νεανική ανεργία αυξάνεται, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι απλά ότι η ανεργία και η φτώχεια έχουν αυξηθεί κατά όρο. Οι αποκλήσεις επίσης μεταξύ των κρατών μελών αυξάνονται και ειδικότερα μεταξύ του πυρήνα και της περιφέρειας της ε, Ευρωζώνης. Και όλα αυτά παρακολύουν ε, το δυναμικό για μια γρήγορη ανάπτυξη του ΑΕΠ. Έχουμε την αιτήσια αναθεώρηση για την απασχόληση που θα δείτε εκεί πολύ αναλυτικά στοιχεία, αλλά θα σας περιγράψω εγώ ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις και προτεραιότητες για την κοινωνική πολιτική, για την πολιτική απασχόληση με βάση την δημοσίευση αυτή και την κοινή έκταση για την απασχόληση που δημοσίευσε στο πλαίσιο της ε, ετήσιας ε, επισκόπησης της απασχόλησης η Κομισιόν. Τον πρώτα απ' όλα στοιχεία της απασχόλησης. Μειώθηκε η απασχόληση και πέρυσι, με εξαίρεση μία μόνο κατηγορία που είναι η πιο μεγάλη ηλικία εργαζόμενη σε ό,τι αφορά τις θέσεις ε, τη κενές. Ε, δεν μειώθηκε πολύ ο αριθμός από το 2010 και μετά, η ανεργία όμω αυξάνεται έκτοτε. Και αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι η έλλειψη ευκαιριών στην αγορά εργασία δεν θα αντιμετωπιστεί αν δεν επενδύσουμε περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο και αν δεν δώσουμε μεγαλύτερη στήριξη ε, στους ανέργους. Οι απώλειες θέσεων εργασίας ε, επίσης δεν ήταν ομοιόμορφα κατανεμημένες ε, και οι ε, υπήκοοι τρίτων χαρών, ε, χωρών, άτομα ε, με επισφαλείς θέση εργασία ή με χαμηλή εξειδίκευση έχουν πληγεί περισσότερο από τους υπόλοιπου. Ο κατακαιρματισμό τη αγορά εργασία παραμένει ένα οξύ πρόβλημα. Το είδαμε και με τα χαμηλά επίπεδα μετακίνηση από πιο επισφαλή σε, λιγότερο επισφαλείς θέση εργασία και με άλλα στοιχεία. Επίσης, η άνθρωποι οι οποίοι ε, είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, ε, παρουσιάζουν κάποια ελαφρά μείωση. Επίσης δεν υπάρχει εξισορρόπηση της ζήτησης και της προσφοράς των δεξιοτήτων. Δεν λαμβάνονται δηλαδή ακόμη ανάγκη, επαρκώ επαρκώς υπόψη οι ανάγκε, η ανταγωνιστικότητα. Πρέπει λοιπόν να εξορροπηθούν αυτές οι ανάγκες και ταυτόχρονα πρέπει να στηριχθεί περισσότερο η ζήτηση εργασίας. Η ζήτηση εργασίας όμως περιορίζεται λόγω των φορολογικών διαφορών που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Η προτινόμενη ανάπτυξη του ΑΕΠΑ ίσως συνοδευτεί με μείωση της ανεργίας και της φτώχειας. Ωστόσο η πρόοδος αυτή πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα είναι βραδία. Δεν θα βελτιωθεί δραστικά η κατάσταση των ανέργων και των φτωχών οικοκυριών παρά μόνο αν δοθεί μεγάλη στήριξη από τις κυβερνήσεις για τις εξελίξεις απασχόλησης και, τα κοινωνικά θέματα έγινε ε, πρόσφατα μία μελέτη η οποία εξετάζει τα στοιχεία αυτά αναλυτικά και μας οδηγεί σε νέα ε, κατεύθυνση στην ανάλυση μας. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι κατά μέσο όρο ένας στους τρεις Ευρωπαίους ε, που ζει στο όριο της φτώχειας καταφέρει να ανεβεί το όριο της φτώχειας ε, μέσα σε ένα χρόνο. Για να βγει από τη φτώχεια ένας ενήλικος συνήθως ε, βέβαια πρέπει να βρει μια θέση εργασίας. Αλλά δεν αρκεί πάντοτε αυτό. Η εξέβρεση θέση εργασίας είναι διέξοδος από τη φτώχεια μόνο στις μισές περιπτώσεις. Πολλά εξαρτώνται από το είδος της δουλειάς, από την αμοιβή και από τις ώρες εργασίας και από τη σύνθεση όμως του νοικοκυριού και την κατάσταση, δηλαδή το αν είναι εργαζόμενος ή όχι ο σύντροφος ή η σύντροφος. Επομένως ε, δεν σημαίνει το ότι βρήκε κάποιο δουλειά ότι αυτόματα έχει φτάσει και σε ένα αξιοπρεπές ε, επίπεδο διαβίωσης και αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις και για το τι μπορεί κανείς να περιμένει από την τρέχουσα οικονομική ανάκαμψη, μείωση της ανεργίας ε, βαθμιαία, δεν θα αρκέσει από μόνη της για να αναστραφεί η τάση ε, αύξηση των ε, επιπέδων φτώχειας, που η φτώχεια θα παραμείνει ένα πρόβλημα αν εξακολουθεί να υπάρξει αυτή η πόλωση μεταξύ χαμηλών και υψηλών μισθών και μερομιστίων και αν αυξηθεί ή παραμείνει στα επίπεδα αυτά η μερική απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν οι χαράκτε πολιτική να δώσουν σημασία και στη δημιουργία θέσεων εργασία, αλλά και στην προσβασιμότητα και το χαρακτήρα, τη φύση των νέων θέσεων εργασία, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μια αλληλέγγυα αγορά εργασία. Μια αγορά σε για όλου. Επίση, η σωδηματική υποστήριξη και άλλα τέτοια μέτρα κοινωνικά θα πρέπει να συνεχιστούν ιδίω για ή μάλλον ακόμη και για τα νοικοκυριά που έχουν μέλη που εργάζονται. Θα ήθελα τώρα, αξιότιμοι ε, βουλευτέ, να σα υπογραμμίσω ορισμένα από τα βασικά πορίσματα του νέου πίνακα επιδόσεων. Εκεί κάναμε μία ανάλυση για πρώτη φορά και κάποιων στοιχείων ε, της κοινή ε, επισκόπησης της απασχόλησης. Για να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτή ο πίνακας επιδόσεων ένα ένα νέο εργαλείο για να εντοπίσουμε τα οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα ή τα προβλήματα απασχόλησης. Πέντε είναι οι βασικοί δείκτες. Η συνολική ανεργία, η νεανική ανεργία και πώς οι νέοι δεν είναι, ανεργια ειναι ανικη απασχόλησης ε, και επιμόρφωσης. Τρίτον, πραγματικές αλλαγές ε, σε ό,τι αφορά το διαθέσιμο εισόδημα. Τέταρτον, ποσοστό του ε, πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο φτώχεια και πέμπτον οι ανισότητες εισοδηματικέ. Αυτός ο πίνακα επιδόσεων δείχνει πόσο επίμονα έχουν διατηρηθεί αυτές οι ανισότητες, ε, ιδιω εντο Ευρωζώνη. Η κοινωνική κατάσταση, η ανεργία στην Νότια Ευρώπη είναι οξύτατη ε, και έχουμε μια βαθιά κρίση στον αυτό. Αλλά ακόμη και πιο ανθεκτικά κράτη-μέλη επηρεάστηκαν μειώθηκε η συνολική ζήτηση, διαβρώθηκε η εμπιστοσύνη. Αυτές οι αποκλήσεις λοιπόν που αυξάνονται φαίνονται ξεκάθαρα στα ποσοστά της ανεργίας, της συνολικής και της νεανικής ανεργίας και των αναγκών των νέων. Μεγαλύτερες αποκλήσεις εντός Ευρωζώνης παρατηρούνται παρά εκτός Ευρωζώνης. Αυτό αφορά και τις ανισότητες και τα, το εισόδημα των οικοκυριών. Τα ποσοστά φτώχειας επίσης έχουν αυξηθεί στην περιφέρεια της Ευρωζώνης ενώ στον πυρήνα παραμένουν σταθερά τα ποσοστά αυτά. Μετά την έγκριση του πίνακα επιδόσεων από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο, πρέπει πλέον τώρα να το αξιοποιήσουμε πλήρω το εργαλείο αυτό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, λαμβάνοντα υπόψη και τι απόψει άλλων εμπλεκομένων φορέων. Εμεί συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα ενταχθεί στο σύστημα τη οικονομική διακυβέρνηση και ιδιαίτερα στην πολυμερή εποπτεία αλλά και στη διατύπωση των συστάσεων αναχώρα. Αξίζουμε βουλευτέ, ολοκληρώνοντα. Θα ήθελα να εστιάσω στι βασικέ προτεραιότητε στον τομέα τον κοινωνικό και τη απασχόλησης για το έτος 2014. Οι προκλήσεις παραμένουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ίδιες με τις περσινές. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακόμα πιο οξύες οι ανάγκες, άρα και οι προτεραιότητες ε, μοιάζουν πολύ με αυτές τις τελευταίες ε, τήσιας επισκόπησης της απασχόλησης. Συμμετοχή στην αγορά ε, εργασίας, θέσεις εργασίας, ε, δημιουργία νέων δηλαδή, σημαντικό. Μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενισχυθούν και με τη μεγαλύτερη στήριξη για τον παναπροσανατολισμό των νέων ανθρώπων σε παραγωγικές δραστηριότητες. Η εγγύηση για την νεολαία. Είναι ένα μόνο παράδειγμα προβλεπτικών πολιτικών απασχόλησης. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα, ιδίως ό,τι αφορά την προώθηση της ζήτησης απασχόλησης, φορολογία, κοινωνικά επιδόματα πρέπει να συνδυαστούν, ιδίως για τους ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα. Βέβαια, αυξάνονται παρά τις ε, τα προβλήματα παρά τις ε, συστάσεις που απευθύνουμε. Για τη δημιουργία θέσεων ε, εργασίας θα πρέπει να προωθηθεί και η ανταγωνιστικότητα, η σχέση κόστους ωφέλους και να υπάρξει περισσότερη ζήτηση. Επίσης έχουμε πληθωριστικές πιέσεις από τους μισθούς, πολύ χαμηλές αυτή τη στιγμή, γι' αυτό υπάρχει περιθώριο με τους μισθούς να αυξηθεί η ζήτηση, ιδίως σε χώρες που τα καταφέρουν καλά. Επίσης, θα πρέπει να επενδύσουμε στη διατήρηση της απασχολησιμότητας και της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού, με ενεργό υποστήριξη, κατάρτιση, επιμόρφωση, ιδίως σε, στην πράσινη οικονομία, στη λευκή ε, οικονομία, στην πράσινη οικονομία. Πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας, όπως και των μακροχρόνιων έργων, των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων, των γυναικών και των, ατήμων, των ατόμων ε, που αποτελούν μετανάστες οικονομικούς. Πρέπει να στηριχθεί επίσης η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας. Πρέπει να βελτιωθούν ε, πρέπει να βελτιωθεί η προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων και εργαζομένων να προωθηθεί κινητικότητα, να προωθηθούν δημόσιες υπηρεσίες. Έχουμε προτάσεις της Κομισιόν πολύ σημαντικές όπως είναι το Γιούρες. Πρέπει να μειωθεί ο κατακαιρματισμός αγοράς εργασίας και των αγορών, αλλά η ασφάλεια των θέσεων εργασίας να είναι ικανή. Και πολλά άλλα μέτρα που ε, θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης ε, και των δεξιοτήτων είναι σημαντικά. Πρέπει να βγούμε πιο ισχυροί από αυτή την κρίση. Θα πρέπει αυτό να γίνει και με τον εξυγχρονισμό των κοινωνικών πολιτικών. Χρειάζονται λοιπόν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ενεργοποίηση και αναβάθμιση των κοινωνικών επενδύσεων. Βέβαια, βελτίωση και του ανθρώπινου κεφαλαίου και της κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτά όμως απαιτείται η επαρκή πρόσβαση και στα κοινωνιακά, προνοιακά επιδόματα και στι κοινωνικέ υπηρεσίε. Τέλο, κυρίε και κύριοι, να υπογραμμίσω την ελπίδα τη Κομισιόν ότι το 2014 το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα χαρακτηριστεί και από τη μεγαλύτερη και πιο ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Και αυτό θα πρέπει να γίνει όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση των διαθετικών μεταρρυθμίσεων και άλλων μέτρων πολιτικής που θα βελτιώσουν την απασχόληση και θα αποκαταστήσουν την κοινωνική πρόοδο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Ο Φίλιπ Ντεμπάκερ, συνάδελφος από την ΕΚΟΝ για την ετήσια έκθεση ανάπτυξη, θα μας κάνει μια παρουσίαση. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για την εισαγωγή σας. Με χαρά σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εισηγητής της έκθεσης για την ε, έκθεση ανάπτυξη του 2014. Αυτό ήθιστε να γίνεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οικονομικών και υποθέσεων και κοινωνικών υποθέσεων. Εξετάζουμε τις προβλέψεις της Επιτροπής, κάτι που είναι το τμήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας που συνεχίζεται και πρέπει να διευκρινιστεί σε κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν τη δημοκρατική λογοδοσία και την ευθύνη που έχουν ε, ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μου ζητήθηκε να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση κάποιων από τα θέματα που υιοθετήσαμε στην Επιτροπή Οικονομικών και Ομισματικών Υποθέσεων για την έκθεση ανάπτυξης για το 2014. Όπως ήδη αναφέρθηκε από πολλούς μιλητές πριν από μένα, είδαμε τα πρώτα δείγματα μιας πολύ ευάλωτης, αργής, ανάπτυ... μικρής και αργής ανάπτυξης. Αυτό τόσο είναι δείγμα αισιοδοξία, διότι οι πολιτικές τη Ευρωπαϊκής Ένωση, τόσο το six όσο και το ΤΟΥΠΑΚ αλλά και οι διαθωτικέ μεταρρυθμίσει που επιβαλήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, μας επιτρέπουν να ξεφύγουμε από τη συζήτηση για το κατά πόσον η Ευρωζώνη θα κατέρε, κράτη θα έπρεπε να φύγουν από την Ευρωζώνη επαναδέθηκαν δηλαδή με την οικονομική και, σταθε... και χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη και αυτό είναι από τα μεγάλα βήματα μπρος που κάναμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλα είναι καλά, ότι όλα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Όχι. Στην έκθεσή μου ε, εντόπισα πολλά ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε. Ένα από τα βασικά είναι το πώς θα ενισχύσουμε την οικονομία πώς θα αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των εθνικών και ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια οικονομία παγκόσμια που μεταβάλλεται συνέχεια. Αυτό θα είναι κρίσιμο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη της οικονομίας. Αφενός, Υπάρχει η συζήτηση βέβαια για το εργασιακό κόστος και η προσαρμογή του εργασιακού κόστους με την παραγωγικότητα. Ένα μέτρο δυνηρό σε πολλά κράτη-μέλη που εντοπίζει ωστόσο τις, ε, την ανάγκη εφαρμογής βιώσιμων διαθροτικών αλλαγών για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο απαιτεί επενδύσεις, επιπρόσθετες επενδύσεις και δημόσιες και ιδιωτικέ στην έρευνα και ανάπτυξη όπως ε, τόνισε ο επίτροπο και στην εκπαίδευση και στα προσόντα. Και νομίζω ότι έχουμε μακρύ δρόμο ακόμα, ούτω ώστε η ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασία να συντονιστεί με τη διαθεσιμότητα με πολύ πιο εύκολο και ε, σωστό τρόπο. Εντοπίσαμε για το ευρωπαϊκό επίπεδο μια βασική προτεραιότητα να δουλέψουμε για την υλοποίηση της την ολοκλήρωση συγγνώμη, της ΟΝΕ. Ε, υπήρξε ένα μεγάλο βήμα μπρος που ήταν η Τραπεζική Ένωση ε, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βοήθησε στη σταθεροποίηση του οικονομικού συστήματος. Αυτό είναι η εφετηρία όμως. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να μπορέσει το τραπεζικό σύστημα να επανασυνδεθεί με τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν ο κατακαιρματισμός που βλέπουμε σήμερα ε, παίζει ρόλο. Η, ενσωμά... ολοκλήρωση της, ε, της χρηματοοικονομικής αγοράς είναι κρίσιμη για την επόμενη θητεία και για την Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο. Όπω ήδη αναφέρθηκε από τον Επίτροπο κύριο Άντορ, Ζήτημα μεγάλο είναι πώ θα εξασφαλίσουμε ότι η αγορά εργασία θα λειτουργεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Όχι μόνο μέσα στα κράτη-μέλη, αλλά και μεταξύ κρατών μελών για να υπάρξει θετική προσέγγιση στη μετανάστευση, στην αποδημία και την εργασιακή κοινωνικότητα γενικότερα στην Ένωση. Βεβαίω, τα κράτη-μέλη έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση που περιλαμβάνει και εντοπίζει η έκθεση. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει η πρόεδρος. Υπάρχει η χρέωση, των, το χρέος των κρατών μελών που αυξήθηκε κατά 90% στο 90% του ΑΕΠ. Αυτό επιβαρύνει την ανάπτυξη. Επίσης, ε, επιβάλλουμε ε, μεγάλο βάρο, μεγάλο άχθο στι μελλοντικέ γενιές. Πώ θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Όπως είπε ήδη ο Επίτροπος κ. Ρεν, υπάρχει αυτή η δημοσιονομική εξυγίανση για την ανάπτυξη. Θα είναι αναγκαίο στο μέλλον το σύστημα να παραμείνει στέρεο Ταυτόχρονα ωστόσο εντοπίσαμε και άλλε προτεραιότητε που πρέπει να, να ακολουθηθούν από τα κράτη-μέλη. Μίλησα για τι βασικέ διαθωτικέ αλλαγέ στι στις αγορές συμπλήρωση μια, ολοκλήρωση μιας σειρά μεταρρυθμίσεων, αντιμετώπιση τη φοροαποφυγής και τη φοροδιαφυγής και το γεγονό ότι σε επίπεδο κράτου μέλους πρέπει να επανασυνδέσουμε την οικονομία με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ενέργεια και εκπαίδευση. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ο κατακαιρματισμό του χρηματοοικονομικού συστήματο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι επιπτώσει αυτού είναι έλλειψη πρόσβαση ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι η σπονδυλική στήλη τη ευρωπαϊκή οικονομία. Αν δεν έχουν πρόσβαση στην ε, πίστη, ε, στην ε, δανειστική πίστη, αυτό είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπιστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κλείνω. Ένας μεγάλος λόγος της διοργάνωσης εκδήλωσή μας είναι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι τα μέτρα είναι δικά μας, τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά. Ταυτόχρονα, ωστόσο, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από την δημοκρατική λογοδοσία. Και η διαδικασία που περιγράφεται στο εξάμεινο, στο six-pack, στο two-pack είναι διαδικασίες νέες και πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την δημοκρατική λογοδοσία της διαδικασίας. Προσβλέπω και άκουσα τα τελευταία λεπτά πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις για το πώς μπορεί να ενισχυθεί αυτή η λογοδοσία η έκθεση μου περιλαμβάνει σαν κρίσιμο στοιχείο τη δημοκρατική λογοδοσία. Αν θέλουμε να πείσουμε του πολίτες μα ότι τα βήματα που λαμβάνονται είναι αναγκαία, οδυνηρά ίσως αλλά αναγκαία για να ξανασυνδέσουμε την οικονομία με την αγορά εργασία και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία τη εκθέσεώς μου. Περιμένω ερωτήσει, ή σχόλια στο γη μέλλον. Ευχαριστώ για ε, την ε, καλή εισήγηση που έχει κάνει. Ε, δίνω το λόγο στον Σέρζο Κουτιέρε, εισηγητή τη Επιτροπή Απασχόληση για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη με τη θερμή παράκληση να μην υπερβεί τον χρόνο των 4 λεπτών, κύριε Κουτιέρες. Ευχαριστώ, καλησπέρα. Σας ε, ζητώ συγγνώμη επειδή όλες οι ομάδες πραγματευόμαστε τις συμβαστικές τροπολογίες της έκθεσης καθυστέρησα. Πρώτα απ' όλα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή καλύτερα που φαίνεται να εστιάζεται η πολιτική συζήτηση στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, για να τα πω απλά, κάποια μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και κάποια κράτη και κάποιοι βουλευτές ε, λένε ότι επανέρχεται η ανάκαμψη και έχουμε κάποια θετικά στοιχεία για να μπορεί να γίνεται λόγος για ανάκαμψη. Όμως άλλοι και μεταξύ αυτών και εγώ, ναι μεν δεν αρνούμεθα κάποια στοιχεία, κάποια σημάδια ανάκαμψης, αλλά θεωρούμε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν για την επίτευξη αυτής της ανάκαμψης οδηγούν σε μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και αποκλείσει στα κράτη-μέλη και εντός των κρατών μελών και μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ πολιτών, για να το πω έτσι πιο εύγλωτα για να μπορεί το τμήμα του κύριου Ρέν να μιλά για ανάκαμψη και να μας ε, αναφέρει όλα αυτά τα θετικά. Έχει θυσιαστεί η πλειοψηφία των κοινωνικών στόχων και στόχων απασχόλησης που είναι αρμοδία του κυρίου Άντορ. Ανεξάρτητα σε ποια πολιτική οικογένεια ανήκουμε, από ποια χώρα προερχόμαστε, πρέπει να λύσουμε τα μακροοικονομικά μας προβλήματα και τα κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα απασχόλησης. Αλλιώς θα επανέλθουν βραχυπρόθεσμα και θα δημιουργήσουν ε, ζητήματα και μακροοικονομικά πολύ σοβαρά. Στην Επιτροπή Απασχόλησης λοιπόν έχουμε βασιστεί σε τέσσερις ιδέες. Αυτή είναι οι άξονες της έκθεσής ε, μας. Πρώτα απ' όλα μια κριτική. Δεν υπάρχει δέσμευση ούτε από τα κράτη-μέλη ούτε από την Κομισιόν ε, απέναντι στις ε, συστάσεις ε, του Κοινοβουλίου και ιδίως αυτές που εγκρίνονται για τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα της απασχόλησης. Κάτι που μας ανησυχεί πάρα πολύ από την έναξη τη όλης διαδικασίας είναι η δημοκρατική νομιμοποίηση που θα πρέπει να αντισταθμίζει τη μεταφορά της εθνικής κυριαρχίας προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτή η δημοκρατική νομιμοποίηση γίνεται με γνωμοδοτήσεις αλλά και με συναπόφαση. Τρεις βασικές μας Πρώτον, στο ευρωπαϊκό επίπεδο να προωθήσουμε διοργανική συμφωνία Κομισιών Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη συναπόφαση. Δεύτερον, να εγγυηθούμε ότι και τα κράτη-μέλη όταν θα εκπονούν τα εθνικά σχέδια μεταρρυθμίσεων αλλά και τα προγράμματα σταθερότητα σύγκληση, θα πρέπει ε, να απευθύνονται πρώτα στα εθνικά κοινοβούλια και μετά να στέλνουν αυτά τα σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίση πρέπει να είναι εγγυημένο και ο κοινωνικό διάλογο. Επίση, θεωρήσαμε σκόπιμο να προτείνουμε πριν τη συνεδριάση του Ευρωπαϊκού Σύμβουλου, όπω γίνεται με το ΕΚΟΦΗΝ, να συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δεύτερη ιδέα. Φοβούμεθα ότι επειδή θα υπάρξουν κάποια θετικά σημάδια, μήπως από αυτό χάσουμε την ανάγκη της ανάκαμψης. Μπορεί η ανάκαμψη να γίνει με βραδύτερους ρυθμούς, να είναι μικρότερη. Και επίσης μπορεί να έχει αποτέλεσμα και την αύξηση ε, κοινωνικών χασμάτων και ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών. Ακόμη και σήμερα ένας στους πέντε νέους είναι άνεργος. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και όσοι βρίσκουν δουλειά συνήθω είναι επισφαλή η θέση εργασία. Υπάρχει κίνδυνο τριπλασιασμού ε, του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυξάνεται ο κοινωνικός αποκλεισμός ε, και τα εισοδήματα, ε, το εισοδηματικό χάσμα αυξάνεται και φαίνεται να χάνεται η μεσαία τάξη. Δεν θα πρέπει να είμαστε ούτε αυτάρισκοι. πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι η στρατηγική μας για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά ή κατά πλειοψηφία στην εσωτερική υποτίμηση του μισθολογικού κόστου για τρει λόγου. Πρώτον, γιατί ε, ο πολίτη αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αδικία μεγάλη για την έξοδο από την κρίση. Χάνουν θέσει ε, δουλειά. Πολλοί. Χάνουν ε, μεγάλο κομμάτι του μισθού του περισσότεροι. Επίση, για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε τι γίνεται και με τις βαθμολογήσεις από τους οίκους αξιολόγησης. Τι μοντέλα οικονομικά και κοινωνικά ε, προωθούνται. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Παραγωγικών Επενδύσεων υπέρ της απασχόλησης και της εργασιακής μεταρρύθμισης με μεγαλύτερη ευελιξία. Ο μισθός να συνδέεται με την παραγωγικότητα, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει η σχέση μεταξύ μεγαλύτερης παραγωγικότητας και καλύτερων εργασιακών συνθήκων. Σήμερα, για παράδειγμα, σε κάποια μέσα επικοινωνία, αναφέρεται ότι προειδοποίησε η Κομισιόν ότι στην Ισπανία δεν είναι εγγυημένο ότι κάποιο έχει δουλειά, βγαίνει και από τη φτώχεια. Και ένα στοιχείο που πρέπει να μα κάνει να σκεφτούμε πολλού σήμερα, όχι μόνο για τι ε, οικονομικέ στρατηγικέ που ακολουθούμε, αλλά και για τι κοινωνικέ επιπτώσει αυτών των στρατηγικών και για το ποιο είναι το κοινωνικό μοντέλο που θέλουμε να υπερασπιστούμε. Τρίτη και τελευταία ιδέα, και επειδή πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι αρνητικέ επιπτώσει. Ε, στην εσωτερική ζήτηση λόγω αυτών των ε, περικοπών στους μισθούς και επειδή εξαρτώμαστε και από την κατάσταση στις τρίτες χώρες, όλα αυτά μας κάνουν να λαμβάνουμε υπόψη μας την ανάγκη για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό ζητούμε μια πολύ πιο φιλόδοξη στρατηγική δημιουργία θέσεων απασχόλησης ιδίως για τους νέους. Καλύτερη χρήση των ε, κοινωνικών ταμείων και των διαφθορτικών ταμείων. Τα κράτη-μέλη να μπορούν να δίνουν ε, περισσότερα κονδύλια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους. Η Ισπανική κυβέρνηση έκανε μια πρόταση να μην υπολογίζεται στο έλλειμμα ε, το κομμάτι των επενδύσεων που πηγαίνει για την ε, απασχόληση των και τρίτον κινητικότητα μεγαλύτερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενίσχυση του έουρες και της φορητότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων γιατί ξέρουμε ότι πολλοί νέοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους και να μεταναστεύσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουτιέρες. Ανοίγουμε τον κύκλο των ερωτήσεων-απαντήσεων. Ε, θα κάνουν ερωτήσεις πρώτα τέσσερις ε, συνάδελφοι. Ε, θα απαντήσουν οι δύο επίτροποι και ανοίγουμε μετά το δεύτερο κύκλο. Ξεκινάμε με τον κύριο Φιλίπ Μαρινή, πρόεδρο της Επιτροπής ε, Οικονομική Γαλλικής Γερουσίας. Madame la Présidente. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ένωση, ε, η, μάλλον η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, κατ' εμένα είναι απογοητευτική. Ναι μεν, αληθεύεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος στις Βρυξέλλες, η συνεδρίαση, μάλλον ε, μεταξύ όλων των επιτροπών αύριο το πρωί θα μας επιτρέψει να πραγματευτούμε συγκεκριμένα ζητήματα και να έχουμε πραγματική ανταλλαγή απόψεων. Όμως πρέπει να ε, συμφωνήσετε ότι διέπεται, διέπονται όλες αυτές οι συνεδριάσεις από τις αρχές του, ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής ορθότητας σε σχέση με το Βίλνιους που τα ταβεί για το προηγούμενο εξάμεινο. Εγώ βλέπω πραγματική όπιστοδρόμηση σε σχέση με το Βίλνιους. Στο Βίλνιους προβλεπόταν η κατάρτιση ενός κανονισμού, η συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας, ώστε να προσδιοριστεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα εθνικά κοινοβούλια. Πώς μπορούν οι βουλευτές πραγματικά να συμμετάσχουν σε κάτι εάν δεν έχουν τη μέση διάταξη στη διάθεσή τους, αν δεν υπάρχει γραμματεία, αν δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιος εισηγητής και αν όλα γίνονται σαν οι πληροφορίες ε, ε, έρχονται από πάνω προς τα κάτω μόνο. Οι ψηφοφόροι μας πολύ συχνά εκφράζουν τα παραπονά τους, ε, ιδίως όταν πλησιάζουν και οι ευρωεκλογές. Και πραγματικά αυτό πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι για εμάς. Σα ζητώ λοιπόν κύριε Επιτρόπε να πάτε πιο μακριά, να εμπιστευτείτε τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί ο ρόλο του είτε το θέλουμε είτε όχι, θα είναι κρίσιμο για την δημιουργία και την εφαρμογή τη Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Κύριε Μαρινή, συμμεριζόμαστε απόλυτα και συμφωνούμε με το συμπέρασμά σα, αλλά θα ήθελα να σα πω παρόλα αυτά ότι το ζήτημα το οποίο θέτεται συζητήθηκε στην προηγούμενη συνεδρία και ανακοινώσαμε ότι η ελληνική προεδρία θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις και το θέμα ε, της διαδικασίας θα ρυθμιστεί εξάπαντος επί Ιταλικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πάντως για την παρέμβασή σας. Το λόγο έχει ο κύριος Αντρέι Γκαλαζεύσκη από την Πολωνική Βουλή. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη και έτσι ενισχύουμε και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα δημοσιονομικά. Κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του. Πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να ενισχύσουμε την πολωνική οικονομία και να προωθήσουμε και την κοινωνική ανάπτυξη. Σημεριζόμαστε όμως και την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάζει συστάσεις. προς τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε επίσης ότι είναι καλή πρακτική να διορθώνονται αυτές οι συστάσεις. Πιστεύουμε ότι έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο οδηγεί σε συζητήσεις ε, στο Πολωνικό Κοινοβούλιο. Οι συζητήσεις αυτές ε, αρχικά ήταν πολύ πολιτικές και συναισθηματικές, ε, τώρα έχουν γίνει πιο ε, ρεαλιστικές, αντικειμενικές. Σε πολλές περιπτώσεις το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο διαφορετικές ε, οικονομικές πολιτικές ε, στην ε, Ευρώπη ε, οδηγεί σε πολύ αργές αντιδράσεις από τα θεσμικά όργανα όσον αφορά την ε, παγκόσμια οικονομία. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με τη κοινή λογική, είσαστε υπέρ των δαπανηρών πηγών ενέργειας σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Από την άλλη, είναι πολύ δύσκολο για τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν την ισορροπία ανάμεσα στις δημόσιες επενδύσεις και στις δημόσιες δαπάνες. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όταν οι οικονομικοί κύκλοι των κρατών μελών εξαρτώνται από την ε, ημερομηνία των κοινοβουλευτικών εκλογών, διότι σε μια προεκλογική περίοδο οι πολιτικοί τείνουν να προβάλλουν λαϊκιστικά συνθήματα και όχι να επικεντρώνονται στις μεταρρυθμίσεις. Μαρτίνες Μποζάλτε από την Ισπανική Βουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ισπανία, μάλλον το Ισπανικό Κοινοβούλιο, υποστηρίζει συμφωνεί απόλυτα και θεωρούμε ότι μας αντιπροσωπεύουν οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί. Στην Ισπανία πιστεύουμε ότι δουλέψαμε σωστά με την Ευρώπη τα δύο αυτά χρόνια, κάτι που μας επέτρεψε να διορθώσουμε την πορεία της ισπανικής οικονομίας. Ωστόσο, θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για προτεραιότητες της Ένωσης, συνήθως μιλάμε για ωραία συμπαθητικά μέτρα που εφαρμόζονται σε όλους. Ωστόσο, πολλές συστάσεις, όχι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά της Επιτροπής, ε, αφορούν μόνο κάποια κράτη. Δεν εφαρμόζονται σε όλα. Όταν βρισκόμαστε στα εθνικά κοινοβούλια, μάλιστα, τα θετικά μέτρα, η κυβέρνηση τα πιστώνει στον εαυτό τη ενώ τα κακά μέτρα συνήθως λέει ότι επιβάλλονται από τις Βρυξέλλε. Και με πολύ ειδικό τρόπο για τη χώρα μας. Αυτό στην, συμβάλλει στην ε, απομάκρυνση του πολίτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό νομίζω, και θέλω να το υπογραμμίσω, ότι είναι πολύ σημαντική επαγρύπνηση της Ένωσης σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών χωρών, διότι αυτό που κάνει ένας, ένα κράτος μπορεί να επηρεάσει όλα. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε και μεταξύ των προτεραιοτήτων πρέπει να εξετάσουμε και να είναι τα μέτρα, μέτρα για όλους, για όλες τις χώρες που εφαρμόζονται σε όλους και που είναι απαιτητά σε όλους, από όλους. Δεν νομίζω ότι συμβάλλει στο κοινοτικό κεκτημένο αγάπης το ότι κάποια φαίνεται, νομίζω πολίτης ότι κάποια κράτη τα μετράμε με διαφορετικό, με, με διαφορετικό μέτρο από ό,τι άλλα. Αυτά και ευχαριστώ. Κύκλο των ομιλητών με τον κύριο Κωνσταντίνο Πουπάκη από το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ξεκάθαρο ότι η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της οικονομικής διακυβέρνησης οι επιπτώσει τη κρίση αλλά και οι πολιτικέ που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση τη διαμορφώνουν μια έκρηθμη κοινωνική κατάσταση στο εσωτερικό τη Ένωση. Έτσι, το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου διευρύνεται επικίνδυνα, οι κοινωνικέ ανισότητε οξύνονται, η ανεργία και η ανεργία των νέων έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, στη χώρα μου η ανεργία των νέων ξεπερνάει και το 57%, η φτώχεια εξαπλώνεται, ήδη ένα στου τρει Έλληνε εμά κινδυνεύουν από φτώχεια. Ταυτόχρονα, και ενώ οι κοινωνικές δαπάνες περικόπτονται συνεχώς, οι χαμηλόμενες διεπομίζονται δυσανάλογα φορολογικά βάρη, είτε με άμεση είτε με έμεση φορολόγηση, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη θέση φορολόγησης φυσικών προσώπων. Τα εισοδήματα περιορίζονται σημαντικά, κυρίως λόγω του βίαιου κατακαιρματισμού των αγορών εργασίας, με δυσμενείς προεκτάσεις για την πραγματική οικονομία και την απασχόληση. Η ίδια η εργασία δεν προστατεύει πια από τη φτώχεια, με του φτωχού εργαζόμενους να πολλαπλασιάζονται επομένως οι μακροοικονομικές πολιτικές δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικές όσο στερούνται κοινωνικού περιεχομένου και αναπτυξιακού προσανατολισμού. απαιτείται λοιπόν ένα ισχυρό κοινωνικό σύμφωνο για την ευρώπη και πρέπει όλοι να το καταλάβουμε με γνώμονα μια ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και σεβασμό στις αξίες του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Σε αυτή την κατεύθυνση και με δεδομένα τα συμπεράσματα της κοινή έκθεσης για την απασχόληση θα ήθελα ρωτήσω πώς πρόκειται να επιτευχθεί φέτος στις ειδικέ αναχώρασης τάσεις η αναγκαία ισορροπία μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής διάστασης και θα υπάρξει ειδική μέρημνα για τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής όπως η Ελλάδα και φέρονται αποκλεισμένα πλήρως από τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020. Ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει ο Επίτροπος κ. Όλη Ρεν. Θα προκαλέσω για μια σύντομη απάντηση όσο μπορείτε στους ερωτώντες. Ε, τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο για να δώσω τη δυνατότητα και στον συνάδελφό μου τον Λάσλο Άντορ για να απαντήσει όσον αφορά την πολιτική της αγοράς εργασία και την κοινωνική πολιτική. Πρόκειται για θέματα πολύ ε, σημαντικά και κεντρικά για το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον των νέων μας. Ο κύριος Καλασεύσκη ανέφερε ότι η Κομισιόν ε, ακούει αυτά που λέγονται. Έχω ακούσει πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε. Ε, εκτιμώ το ότι αντιμετωπίζετε με τόση σοβαρότητα τα θέματα αυτά. Να αναφερθώ στην παρέμβαση του Φίλιπ Τεπάκερ, ο οποίος ε, ανέφερε κάποια πολύ σημαντικά θέματα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και για την απασχόληση για την ε, κοινωνική ε, ευημερία μας. Περιγράφει στην έκθεσή του τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Τονίζει τη σημασία της ελεύθερης κινητικότητας στην αγορά εργασίας και θεωρεί λυπηρό ότι επηρεαζόμαστε σε διαφορετικό βαθμό από τις ε, χρηματοοικονομικές αγορές ε, στις διαφορές χώρες της Ευρώπης. Θα πρέπει να εξαλείψουμε τα εμπόδια στην ανάπτυξη που υπάρχουν, μεταξύ άλλων, δημιουργώντας ε, μια τραπεζική ένωση να δημιουργήσουμε έναν αξιόπιστο και σταθερό τραπεζικό τομέα που να μπορεί να δανείζει στον πραγματικό τομέα της οικονομίας, ώστε να μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη και απασχόληση. Ο κύριος ε, Μαρίνη σχολίασε κυρίως ε, τις μεθόδους εργασίας και αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν επίσης δικαίωμα να προσκαλούν σε ακρόαση τους ε, επιτρόπους στο πλαίσιο της, ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και χαίρομαι που έχω επισκεφτεί αρκετά ε, εθνικά ευρωπαϊκά κοινοβούλια για να παρουσιάσω τα σχέδια μας. Ο κύριος Πουπάκης έχει απολύτως δίκιο ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στις συστάσεις αναφόρα. Αυτό συμβαίνει στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. όπου πραγματοποιείται η ετήσια εποπτεία. Είναι λοιπόν σημαντική η συζήτηση αν οι ε, διάφορες χώρες έχουν εφαρμόσει τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να εξετάσουμε τους εθνικούς στόχους και να τονίσουμε τα μέτρα που δημιουργούν ανάπτυξη και ε, απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ και δίνω τον λόγο στον κύριο Αντόρ. Ε, η σειρά σας για τρία λεφτά επίση. Uh, Ευχαριστώ. Τι να πω σε τρία λεπτά. Να σταθώ σε δύο-τρία σημεία. Πρώτον, είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ αρκετά. Φιλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ολλανδία και τις επόμενες εβδομάδες θα πάω και στο Bundestag καθώς και στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Οι συζητήσεις σε όλα αυτά τα βήματα επέτρεψαν μια πολύ καλή συζήτηση για την κατάσταση σε ένα χώρα, αξιολόγηση και ανάδραση των απόψεων που ακούμε και αυτός ο διάλογος είναι πολύ σημαντικός. Όταν όταν δείτε μάλλον τη συστάσεις σε ένα χώρα πέρυσι, αλλά και όταν δείτε αργότερα τον επόμενο κύκλο συστάσεων θα δείτε ότι προσπαθούμε να κόψουμε και να ράψουμε την ανάλυση και τις ε, συστάσεις ανάλογα με την πραγματική επιτόπια κατάσταση. Η εγγύηση νέων, για παράδειγμα, που το ανέφερε και ο Σγκουτιέρες, ε, είναι ένα σημαντικό εργαλείο, βασίζεται στο επίπεδο της ανεργίας των νέων και των αναγκών των νέων σε μια συγκεκριμένη χώρα και στηρίζεται στην υφιστάμενη εμπειρία κάποιων χωρών ε, για την υποστήριξη της ανεργίας των νέων χρησιμοποιώντας, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία της Ένωσης. Αυτό περιλαμβανόταν στον τελευταίο κύκλο. Θα επανέλθουμε αργότερα φέτος, αξιολογώντας τα προγράμματα εφαρμογής των εγγυήσεων νέων που έχουν συμπληρώσει όλες σχεδόν οι χώρες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ε, νέα πρωτοβουλία ενίσχυσης των νέων. Επίσης, χώρες με, μεγάλο, με σχετικά μεγάλο πληθυσμό Ρωμά έλαβαν πέρσι για πρώτη φορά ειδικέ συστάσεις γιατί ήταν σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι υπήρχε και πολιτική υποστήριξη και ενθάρρυνση στην πρόθεση προγραμμάτων ένταξης που επίσης μπορούν να υποστηριχθούν από τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της Ένωσης. Όχι μόνο το Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτά τα προγράμματα πιστεύω θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της στόχης. Ευχαριστώ. Ε, πανερχόμαστε στον κύκλο των ε, ερωτήσεων από τους βουλευτές και ευρωβουλευτές με την κυρία Ανούς Κασούτα από την Άνω Βουλή Ολλανδίας. Για δύο λεπτά υπενθυμίζω. Dear um, Πρόεδρε, μιλώ ως εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο της ε, Βουλής της Ολλανδίας εμείς ως εκπρόσωποι της Ολλανδίας θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κοινοβουλευτική διάσκεψη για να μοιραστούμε τις βέλτιες, τις, τις πρακτικές με τα κράτη-μέλη και όχι να συζητούμε διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Ολλανδία πήρε μία σύσταση να μεταρρυθμίσει το συνταξιοδοτικό της. Έχουμε μια παλιά παράδοση αποταμίευσης για ιδιωτικές συντάξεις και ξέρουμε ότι η σύνταξη πρέπει να είναι βιώσιμη. Αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία συνδέουμε την ε, συνταξιοδοτική ηλικία με το προσδόκιμο ζωή σιγά σιγά ε, από τα 60 προς τα πάνω. Ο κόσμος έχει αρχίσει ήδη να πληρώνει περισσότερο για τα αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε την διαγενειακή ελεγγύη, τους, ώστε οι νέοι να μπορούν να συστήσουν ένα συνταξιοδοτικό ε, κεφάλαιο. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Άντρο τι πιστεύει για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την γύρανση του πληθυσμού και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε συντάξεις για τα, για τα παιδιά και τα, εγγόνα, και τα εγγόνια μας. Ως εισηγήτρια τώρα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θέλω να ζητήσω από το όλους τους συναδέλφους να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία της συνάντησης για να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε και να αγωνιστούμε για κοινέ λύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφωνού, πρόεδρος. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε φαίνεται ο δικός χάρτης, ένα θεματολόγιο με πολύ λίγη φιλοδοξία. Γιατί για να βγούμε από την κρίση είχαμε κάποια στοιχεία ε, στατιστικά για το 12 που δεν συνδυάζονται όμως με την πραγματική οικονομία και την ανάπτυξη. Είναι πολύ λίγο φιλόδοξα λοιπόν αυτά που λέμε. Δύο σημαντικά θέματα. Ζήτηση προσφορά. Για τη ζήτηση, η φορολογική μεταρρύθμιση, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής της απάτης, ε, της φοροαποφυγής. Πολύ σημαντικό για τη σταθεροποίηση του χρέους και του έλλειμου και για τη χρηματοδότηση της βιωσιμότητας του κράτου πρόνοιας. Το 2014 κατεμένει είναι ένα έτος πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να αναθεωρηθούν, να επικαιροποιηθούν. Υπάρχει και η εξέλιξη στις Ηνωμένε Πολιτείε με τα μέτρα που προτείνει ο Ομπάμα, με τις εξελίξεις και σε επίπεδο όσα. Αλλά εμείς ε, νομίζω ότι ε, λίγο προβλεπτικά μέτρα προωθούμε. Παραδείγματος χάρη έχει καθυστερήσει η οδηγία για την ε, φορολόγηση των αποταμίευσεων. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το έτος 2014. Πρέπει να θεωρηθεί αυτή η οδηγία, η οδηγία για τις θηγατρικές, για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και μια πρώτη οδηγία για τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας που πρέπει να έλθει αυτό το έτος. Λίγη είναι η φιλοδοξία λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι πολύ σημαντικό όμως για την ευρωπαϊκή κοινωνία θα ήταν αυτό. Δεύτερον, έρχομαι στο σκέλος της προσφοράς. Δεν φτάνουν τα χρήματα πράγματα, πράγματι από τις τράπεζες στις επιχειρήσεις, δηλαδή στην πραγματική οικονομία. Κύριε Επίτροπε, τι φταίει. Μήπως ο σχεδιασμός των πολιτικών, της νομισματικής πολιτικής, που δεν είναι σωστός. Δεν δίνονται κίνητρα, δεν ε, παρακινούνται, οι τράπεζες το κάνουν. Τι αλλαγέ πρέπει να γίνουν στην νομισματική πολιτική ώστε πραγματικά τα χρήματα να πηγαίνουν και να φθάνουν από τι τράπεζε στην πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Ντανιέλο Ρουά από τη Γαλλική Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο κύριο Άντορ και τον εισηγητή, διότι η κοινωνική διάσταση πρέπει να υπάρχει σε όλο το εξάμεινο, όχι μόνο στην ετήσια εξέταση της έκθεσης για την ανάπτυξη. Και επιτρέψτε να σας πω ότι η Γαλλική Εθνοσυνέλευση χαίρεται ιδιαίτερα όταν οι επίτροποι ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις της, κάτι δεν είχε συμβεί ποτέ, με τον κύριο Όλι Ρέν το, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να χρησιμοποιήσουν το scoreboard ως εργαλείο ανάλυσης, όχι μόνο ως ένα εργαλείο ορισμού οικονομικών πολιτικών. Θα ήταν σκόπιμο οι συστάσεις να αναχώρα να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομική πολιτική και να λαμβάνουν υπόψη και την ποιότητα της απασχόλησης, την κατάρτιση, την πρόσβαση στην μαθητεία βίου, και την αντιμετώπιση της φτώχειας. Βεβαίως, επιτρέψτε να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί φτωχοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία και σε χώρες που σήμερα φαίνεται ότι τα πάνε καλά. Η φτώχεια αυξάνει παντού. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τα μέσα να την αναλύσουμε ακόμα και μακροοικονομικά. Για την πρόταση της Επιτροπής πρέπει να συμπληρώσουμε τους κοινωνικούς δείκτες. Η πρόταση του εισηγητή κ. Κουτιέρες που θέλει να συμπεριλάβει δίκτες φτώχειας των παιδιών, δείκτη αξιοπρεπούς ε, ε, ε ζωής ε, βιώσιμου μισθού είναι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζουμε τις ε, προτάσεις και επιτρέπουμε να μειώσουμε τις ανισότητες εισοδήματος που δεν εμφανίζονται αυτή τη στιγμή από, τους από τις φυστάμενους δείκτες. Οι κοινωνικοί δείκτες δεν πρέπει να έχουν και δεσμευτικό χαρακτήρα. Οι προτεραιότητες για το εξάμεινο του 2014 θα πρέπει βεβαίω να είναι η ανάπτυξη όπως προτείνει η Επιτροπή, αλλά ταυτόχρονα και η απασχόληση. Αυτό το δείχνει η τεράστια ιστορική πια ε, αρνεργία στη χώρα. Ένας νέος στους πέντε είναι, σε, είναι άνεργος στην Ένωση. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της εξυγίανσης των δημοσιονομικών πολιτικών και της πρόθεσης της ανάπτυξης, στηριζόμενη στις συστάσεις του ΟΣΑ και του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, που επαναλαμβάνω, αμφισβητούν την ταχύτατη προσαρμογή που δέχτηκε η Επιτροπή. Θα πρέπει να το καταλάβει αυτό η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα μιλήσω για την Κροατία, παρότι το πρόβλημα που θα αναφέρω δεν αφορά μόνο την Κροατία. Η Κροατία λοιπόν πρόκειται να ξεκινήσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, θα γίνει μια εσβάθος ανάλυση ως αποτέλεσμα της διαδικασίας για τις ε, μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες. Η Κροατία, όπως οι περισσότερες χώρες, πρέπει να εξυγχρονίσει τη διοίκηση και την οικονομία της. Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να αναθεωρήσει την αγορά εργασίας και όλα αυτά στοιχίζουν. Τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης συνδέονται με τις περικοπές σε επενδύσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει τη στιγμή που οι αναλύσεις δείχνουν ότι περαιτέρω μειώσει μισθών θα οδηγήσουν σε διαφυγή εγκεφάλων και μειωμένο διοικητικό δυναμικό, μειωμένη ανταγωνιστικότητα επίσης, ενώ αυτή θα πρέπει να αυξηθεί. Η ανάλυση επίσης δείχνει ότι οι χαμηλότερες συντάξεις θα οδηγήσουν σε αύξηση της φτώχειας που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 32,7%. Θα η αύξηση του φορολογικού βάρους θα σταματήσει τελείως τις οικονομικές δραστηριότητε. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε την εξή λύση. Τα κράτη-μέλη που βρίσκονται κάτω από το 75% του μέσου ΑΕΠ και που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος θα πρέπει να επιτρέπεται να αφαιρέσουν από τους υπολογισμούς για το έλλειμμα όλες ε, τις επενδύσεις για προγράμματα ανάπτυξης τα οποία συγχρωματοδοτούνται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα επιτρέπεται τουλάχιστον για τα πρώτα λίγα χρόνια, διότι αυτές οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για να προωθήσουν την ανάπτυξη, ε, ενώ η ανάπτυξη ε, μειώνεται διαφορετικά. Ευχαριστώ. Κύριος Ευχαριστώ τον κύριο Ρεν και τον κύριο Άντων. Επιτρέψτε με ένα σχόλιο για αυτό που είπε η Ολλανδή συνάδελφος πριν από λίγο. Η Ουγγαρία πρόσφατα υιοθέτησε μια εθνική στρατηγική ανάπτυξη και προχώρησε σε μια σειρά σοβαρών προσπαθειών που είχαν κόστους αλλά αύξησαν την σταθερότητα της χώρας. Είναι σταθερότερη τώρα η εμπορία από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και θέλω να δώσω έμφαση στην στρατηγική στην εθνική στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξης που καλύπτει όλους τους τομείς μέχρι το 2015 με τρόπο που επιτρέπει την σταθερότητα της χώρας. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα τα μέτρα που έχει λάβει η χώρα, αύξηση των μισθών των ε, δασκάλων, για παράδειγμα, αύξηση μισθών στην ε, μέρη στη βοήθεια στο σπίτι, στο βαθμό βελτίωση στο βαθμό στο ποσοστό προσχώρηση και επαγγελματική κατάρτιση αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται ωστόσο χρόνο. Και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζονται χρόνο για να υλοποιηθούν όλα αυτά και τα αποτελέσματα θέλουν ακόμα περισσότερο χρόνο. Όταν έρθουν στο τα αποτελέσματα, διαπιστώνουμε ότι το ήρθε η ώρα η Ένωση να αυξήσει τις προσπάθειές της υποστηρίζοντας τα, την ολοκλήρωση των νέων αυτών αποτελεσμάτων. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα των εγγυήσεων αυτών ε, είναι βιώσιμο. Ελπίζω να έχουμε μια σταθερότητα στο μέλλον. Η επόμενη πρόκληση θα είναι η χρήση των κονδυλίων της Ένωσης στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Οι τομείς αυτοί είναι τομείς όπου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν μεγάλη έμφαση, γιατί χρειάζεται να βελτιωθεί η συνθήκη, να βελτιωθούν οι συνθήκες για τη μεσαία τάξη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Άλμπα. Είμαι σκιώδης ηγητής ε, του ΕΛΚΑ στην έκθεση για την ετήσια ανάπτυξη. Το πρώτο που πρέπει να πω είναι να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεμπάκερ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του ως προς την ε, σημασία να χρηματοδοτούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ε, παγιωθεί η έξοδος από την κρίση, όπως αναφέρθηκε ήδη. Έχει απόλυτα την υποστήριξή μου σχετικά. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κ. η συγκεκριτή της Επιτροπής Απασχόλησης, νομίζω ότι κανείς δεν είναι ικανοποιημένο με την κατάσταση που βιώνουμε. Βέβαια, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι από τα θετικά στοιχεία που έχουμε. Ωστόσο, πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Νομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο να πούμε στους πολίτες ότι η έξοδος προς την κρίση, από την κρίση θα έρθει από έναν από τους λόγους που μας οδήγησε στην κρίση που είναι περισσότερες κρατικές δαπάνες. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Αντίθετα, χαίρο με αυτά που είπε ο κ. Γκουτιέρες για την εγγύηση για τους νέους και την κινητικότητα. Θα ήθελα να πω στον επίτροπο κύριο Άντορ που το είπε ε, που το είπα σε προηγούμενες ευκαιρίες ότι ε, η δουλειά που κάνει για την εγγύηση νέων είναι πολύ καλή. Να ζητήσω ωστόσο εκ νέου αν γίνεται να φτάσουν τα κονδύλια το συντομότερο δυνατό. Το ζητάνε οι πολίτες. Έχουμε σημαντικότατες εκλογές για την Ευρώπη σε λίγες εβδομάδες. Κάναμε, δημιουργήσαμε τεράστιες προσδοκίες ε, για την εγγύηση νέων. Τώρα ήρθε η ώρα να, εφαρμόσουμε τις, να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας. Εάν δεν έρθουν τα κονδύλια, τι προσδοκίες να υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Μαγντάιρ, για δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριε κυρία Μαγντάιρ, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα απλά να αναφερθώ ειδικότερα στο ρόλο των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει διαμακρό στην Επιτροπή απασχόληση, στην οποία είμαι και μέλος. Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε το, ότι το 85% των νέων θέσεων εργασίας συνολικά στην Ευρώπη προέρχονται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Επομένω. συγκεκριμένα θέτω το εξή ερώτημα ο Επίτροπο Άντορ αλλά και ο Επίτροπο Ρεν, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τι μικρέ επιχειρήσει να δημιουργήσουν νέε θέσει. Επίση, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει την μερική απασχόληση να την στιγματίζουμε, ε, να τη δίνουμε μια αρνητική χρειά. Γιατί και εγώ ως εργοδότρια είδα ότι ο τρόπος ε, να γυρίσουν πίσω οι γυναίκε σε μια ε, δουλειά είναι ακριβώ με μερική απασχόληση. Και δεν χρειάζεται να είναι κάτι χαμηλή εξειδικεύση. Μπορεί να είναι και με πολλέ ε, εξουσίε. Δεν πρέπει να λέμε λοιπόν ότι είναι κακέ αυτέ οι δουλειέ τη μερική απασχόληση. Ε, και την αυτοαπασχόληση ε, είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον αν κανεί δει και την ανεργία των νέων πολύ λίγα κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τους νέους να γίνουν επιχειρηματίες. Αυτό απασχολούμε. Έχουμε το πρόγραμμα Εράσμου για νέους επιχειρηματίες στην Ευρώπη. Διερωτώμε όμω τι άλλο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τους νέους να γίνουν επιχειρηματίες. Τελευταία ερωτώσα είναι η κυρία Χολμάγερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Συνάδελφοι, έχω την εξή ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Διάβασα προσεκτικά τις εκθέσεις και ήταν να υπάρχει μια σημαντική αντίφαση. Από τη μία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί όλο και περισσότερη εκπαίδευση, εξειδίκευση. Από την άλλη όταν ε, μιλάμε για την ε, δημιουργία επιχειρήσεων, ε, μιλάμε για όλο και λιγότερη εκπαίδευση, ότι αυτό θεωρείται εμπόδιο στην εσωτερική αγορά. Εάν δούμε το ποσοστό επιβίωσης των επιχειρήσεων, διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που απαιτούν εξειδίκευση επιβιώνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ όσοι πηγαίνουν, όσοι μπαίνουν στην αγορά με καμία ρύθμιση επιβιώνουν ε, ένα-δύο χρόνια. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ε, να προσφέρει σταθερές ε, και βιώσιμες θέσεις εργασίας και όχι επιχειρηματική ζωή ενός-δύο ετών και μόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε εξειδικευμένους επιχειρηματίες ε, και να μην εφαρμόζουμε απλά μέτρα διακοσμητικά για επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν ένα-δύο χρόνια. Στην ε, Γερμανία έχουμε σχετικό πιστοποιητικό και στην ε, Γαλλία, στις χώρες του Βορρά επίσης υπάρχει, υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις ενώ έχουν οι νότιες χώρες που ακριβώς ε, δεν ε, απαιτούν κάτι τέτοιο από τους νέους επιχειρηματίες. Ε. αλλά οι επιχειρήσεις αυτές επιβιώνουν το πολύ ένα-δύο χρόνια και η ανεργία των νέων ανέρχεται σε 30, 40, 50%. Θέλουμε λοιπόν βιώσιμες επιχειρήσεις Μήπως μπορεί η Κομισιόν να συντονίσει τις εσωτερικές της εργασίες, να γίνει συντονισμός μεταξύ των ε, επιτρόπων, διότι φαίνονται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές από τη μία γενική διεύθυνση στην άλλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χολμάγερ. Προτού να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Ρεν και τον ε, Επίτροπο Άντορ για τις ε, τελικές τους παρατηρήσεις, θα ήθελα πολύ σύντομα να θέσω ένα ερώτημα. προς και τους δύο. Κύριε Αντιπρόεδρε Ρεν, χθες και σήμερα είχαμε συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων προσαρμογής στις χώρες των προγραμμάτων αυτών. Μιλήσαμε και για την εφαρμογή του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και υπάρχει μια λέξη κλειδί που ε, ε, επανεμφανίζεται. Πρόκειται για τη λέξη οικειοποίηση, αίσθημα ιδιοκτησίας αυτό το αίσθημα οικειοποίησης ε, δεν μπορεί να επιβληθεί, πρέπει να επιτευχθεί. Κάτι που απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία. Φτάνω λοιπόν στην ερώτησή μου. Πιστεύω ότι αποκλείοντας ε, τις χώρες των προγραμμάτων από τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου υπονομεύουμε την διαφάνεια και δημιουργούμε δύο κατηγορίες κρατών μελών αυτών που συμμετέχουν στη διαδικασία και αυτών που αποκλείονται από τη διαδικασία. Εξηγήσατε ότι αυτή είναι μια απόφαση που λαμβάνεται στο πλαίσιο της, νομοθεσίας, ε, της δέσμης των δύο νομοθετικών μέτρων του ΤΟΥΠΑΚ. Πιστεύω ωστόσο ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τις αποφάσεις που έχουμε λάβει στο παρελθόν. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μου ερώτηση και η δεύτερη είναι η εξή. Τον περασμένο Δεκέμβριο το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για τους μετρήσιμους στόχους για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Και ε, έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν να σκεφτεί εάν αυτοί οι μετρήσιμοι στόχοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον ε, πίνακα αποτελεσμάτων για τις μακροπρόθεσμες ανισορροπίες. Αυτό είναι κάτι που σχετίζεται και με την έκθεση Πέκερ Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη θέση σας πάνω σε αυτό και η κύριε Επίτροπε Άντορ. Είμαι βέβαιη ότι υπάρχει μια εναλλακτική ετήσια έκθεση ανάπτυξης ε, που έχει προετοιμαστεί από εμπειρογνώμονες που επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θα απαιτηθούν 10 χρόνια ώστε η Ευρώπη να επανέλθει στα ποσοστά απασχόλησης του 2007. Πιστεύω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι πολύ ανησυχητική η πρόβλεψη αυτή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν συμμερίζεστε τη θέση αυτή και να σας ρωτήσω τι πρέπει να γίνει για να αντιστραφεί αυτή η τάση, η οποία σαφώς υπονομεύει την συνεκτικότητα του ευρωπαϊκού έργου στο σύνολό του. Κύριε Ρεν, έχετε το λόγο. Thank you, Vice President. Ευχαριστώ κύριε Ποδηματά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Τι? να απαντήσω με τη σειρά των ερωτήσεων. Συντάξεις. Θα ξεκινήσω με, τους ε, εκπροσώπους των, ε, με τον εκπρόσωπο των κάτω χωρών που ρώτησε σχετικά με την βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων που αφορούν τις συντάξεις. Ε, και μίλησε και για τη σημασία της πραγματικής οικονομίας. Πιστεύω ότι Οι, οι δημογραφικές εξελίξεις αποτελούν σημαντική πρόκληση στις περισσότερες χώρες και μπορώ να σας πω ότι όταν εξετάσαμε πόσα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν λάβει απόφαση σχετικά με μεταρρυθμίσεις της συντάξης, διαθροτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συντάξεων, διαπιστώσαμε ότι 19 από τα 22 τότε κράτη-μέλη. Η εξέταση αυτή έγινε πριν προσχωρήσει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μου δείχνει ότι υπάρχει ένα κύμα μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. όσον αφορά την ερώτηση Σάρο Γκαρσία, πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη ζήτηση. Αυτό είναι σημαντικό ερώτημα. Οι καλές φορολογικές μεταρρυθμίσεις είναι κεντρική σημασία στο πλαίσιο αυτό. Κυρία Αρουά, από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ρωτήσατε επίσης σχετικά με τα θέματα αυτά και θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα πριν σχετικά με την δίκαιη και σωστή φορολόγηση. Θα πρέπει πάντα να αξίζει τον κόπο να εργάζεται κανείς και δεν είναι βιώσιμη λύση το να αφήσουμε μεγάλα χρέη στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε την ε, σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών. Επίσης κύριε Δουά, αναφερθήκατε στην μη συμμετοχή μου στις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης. Ίσως δεν κατάλαβα καλά ή ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι μετά τις συστάσεις μας είχαμε τάσχει σε κοινή συνάντηση των επιτροπών προϋπολογισμού και εξωτερικών της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας μια σοβαρή συζήτηση υπό την προεδρία της κυρίας Γκυγκού. Μπορεί να επανέλθω στο πλαίσιο των επόμενων συστάσεων της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ιδίως υπό το φως του ότι υπάρχουν σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, εξέλιξη ή υποδιαμόρφωση στη Γαλλία τους επόμενους μήνες. Με χαρά λοιπόν θα συμμετάσχω, πάντα χαίρομαι να μετέχω και να έρθω εκ νέου σε συναντήσεις της Εθνοσυνέλευσης. Αν με καλείτε βέβαια ακόμα. Ο κ. Ζάρπα αναφέρθηκε στην ετήσια έκθεση ανάπτυξη του 2014 και τη σημασία τη ρευστότητα προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είπατε ότι ο κ. Δεμπάκερ έχει την υποστήριξή σα στο θέμα αυτό. Συμφωνώ. Και τη δική μου υποστήριξη έχει. Α δουλέψουμε μαζί και α επιτρέψουμε να αρχίσει να ρέει η χρηματοδότηση στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ιδίω στην Νότια Ευρώπη, αλλά κατά πάσα και σε ολόκληρη την Ήπειρο. Και εδώ πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη μαζί και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο των ανεξάρτητων αποφάσεων που λαμβάνει. Πώς θα επισκευάσουμε τον μηχανισμό μετάδοσης ε, της νομισματικής πολιτικής ε, και πώς θα εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για την Ευρώπη. Αυτό είναι σημαντικό γιατί η οικονομική ιστορία δεν γνωρίζει κατάσταση που να υπάρχει ανάπτυξη οικονομική χωρίς αύξηση του δανεισμού. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Η κυρία Μακιντάρη αναφέρθηκε επίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είπε ποιες είναι οι προτεραιότητες της ετήσιας έκθεσης ανάπτυξης. Συνοψίζω, να δημιουργήσουν τους ε, τις σωστές προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις, να, μειώσουν να μειωθεί η γραφειοκρατία, να απελευθερωθεί το επιχειρηματικό δυναμικό, να επιτρέψουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να ενδυναμωθούν με επαρκή προσόντα της αγοράς εργασίας, ένα σημαντικό θέμα. Και τέλος, να υποστηρίξουμε την καινοτομία και την εφαρμογή υλοποίηση κέντρων καινοτομία, αλλά και την πρόσβαση των μικρομεσαίων στην χρηματοδότηση. Νομίζω ότι αυτά είναι κρίσιμα, όπως και αυτά που τόνισε η κυρία Χολμάγερ για την δυνατότητα ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην Ευρώπη πιστεύω δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Έχουμε αρκετές επιχειρήσεις που δημιουργούνται, ωστόσο το επόμενο βήμα, η ανάπτυξή τους, είναι δυσκολότερο από ό,τι για παράδειγμα στις ΗΠΑ, όπου συχνά ο συνδυασμός προβλημάτων στην πρόσβαση στη χρηματοδιοδότηση και η κατακαιρματισμένη ευρωπαϊκή αγορά στην ψηφιακή, στις ψηφιακές υπηρεσίες για παράδειγμα δημιουργεί συμφόρηση σε κάποια σημεία ανάπτυξης. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών, στον τομέα των ψηφιακών ε, υπηρεσιών, για τη βελτίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητα θα είναι ένα καλό εργαλείο για να παρασκευθεί χρηματοδότηση όχι μόνο για το ξεκίνημα αλλά και για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τόσο ώστε να έχουμε στην Ευρώπη μελλοντικούς πρωταθλητές τύπου Google ή άλλων που δημιουργήθηκαν στη ΣΥΠΑ τα τελευταία χρόνια. Περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Τέλος, η κυρία Αντιπρόεδρος, η κυρία μίλησε για την ανάγκη να μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και οι χώρες του εξαμήνου, του προγράμματος, συγγνώμη. Καταγράφω το σχόλιο σας Καταγράφω απόλυτα θα έλεγα το σχόλιο σας και είμαι έτοιμη να, έτοιμος να σκεφτώ πώς θα συνδυάσουμε καλύτερα την παραδοσιακή οικονομική πολιτική με τον συντονισμό με τα προγράμματα που κάνουμε με τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα εξυγίανσης στο πλαίσιο των, της, πρόσφατας, της πρόσφατης νομοθεσίας για το ΤΟΥΠΑΚ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι το να αποδέχεσαι, το να καταλαβαίνεις ότι είναι δικά σου τα μέτρα, είναι κρίσιμο χαρακτήρα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η νέα οικονομική διακυβέρνηση δεν αφορά κυρώσει αλλά συνεργασία, εταιρική σχέση μεταξύ επιτροπή και ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Θέλω να συνεργαστώ, να δουλέψω σε συνεργασία και με τις κυβερνήσεις και με τα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών, γιατί αυτό είναι ο τρόπος για να αυξηθεί το αίσθημα ιδιοκτησίας ε, των μέτρων και να υπάρξουν τα θεμέλια βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασία στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για τις πολλές ε, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Προσβλέπω σε μελλοντική συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Αντιπρόεδρε της Κομισιόν. Τώρα το λόγιο Επιτρόπος Άντορ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, να ξεκινήσω πρώτα στο δικό σας ερώτημα σε σχέση με τη λεγόμενη εναλλακτική αιτήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος Όλη Ρέν, ο οποίος ε, συμμετείχε σε μια συζήτηση για το έγκρο αυτό, ε, θα μπορούσε να απαντήσει, αλλά θα σας πω και εγώ τις δικές μου απόψεις. Εν καιρό κρίσης, όταν ενίοτε ε, η δυναμική της ύφεση, της ανάκαμψης είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, είναι και πολύ δύσκολο βέβαια να δει κανείς πώς ε, όλα αυτά σχετίζονται με τους μακροπρόθεσμους στόχους που εμείς είχαμε καταρτήσει το 2010. Όμως ε, αυτό δεν το συνειδητοποίησαμε μόνο τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, ότι δηλαδή κάποιοι δείκτες πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση, δηλαδή να μην έχουμε πρόοδο, αλλά τελικά απώλεια σε ό,τι αφορά τα επίπεδα της απασχόλησης, και φτώχεια που αυξάνεται σε αρκετές χώρες. Η δική μας προσέγγιση την τελευταία διετία ήταν η εξής. Προσπαθήσαμε να βρούμε νέα εργαλεία και όχι να χαμηλώσουμε τις φιλοδοξίες μας. Αν πούμε ότι το πρόγραμμα ε, που είναι σε μία από τις ε, βασικές ε, πρωτοβουλίες της Κομισιόν αντιμετώπισε προβλήματα λόγω αποκλήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να βρούμε νέα εργαλεία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γυρίσουμε στο σωστό δρόμο, στο σωστό μονοπάτι. Τα εργαλεία ε, τα οποία έχουμε επιλέξει. Το κατά πόσο είναι επαρκή θα το δούμε στο μέλλον. Η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τον απολογισμό, παρέχει μια ανάλυση και κάνει μια έτσι, εξέταση της ε, προόδου των πεπραγμένων, αλλά και η επερχόμενη Επιτροπή του χρόνου θα έχει τη δυνατότητα να καταλήξει σε πιο πρακτικά συμπεράσματα, σε ένα είδος μεσοπρόθεσμης ε, αξιολόγησης αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουν τη διαφορά αυτά τα μέτρα, όπως η για την νεολαία. Ο κύριος ε, Ζάλμπα το ανέφερε αυτό το εργαλείο. Για να κάνει τη διαφορά γρήγορα όμως αυτό το εργαλείο θα πρέπει να υπάρχει και ταμιακή ροή, να ε, διατεθούν τα κονδύλια το συντομότερο δυνατό. Και μετά την, ε, τα σχέδια τα εφαρμοστικά θα πρέπει να έχουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα της πρωτοβουλίας ε, για την νεολαία 6 δις επιπλέον των κονδύλων του Κοινωνικού Ταμείου και βέβαια ο νέος προπολογισμό που πρέπει να δαπανηθεί βέβαια, αλλά πρέπει να σας πω επίσης ότι στις περισσότερες χώρες έχουμε πόρους από την ε, προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού που μόλις ολοκληρώθηκε και που δεν έχουν ακόμη διατεθεί Έχουμε κάποια ποσοστά τη ταξη 65 65-66%. Τα είδαμε με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού χθε. Ελπίζουμε ότι με τα κονδύλια αυτά θα στηριχθούν προγράμματα που προωθούν την απασχόληση των νέων. Η προσπάθειά μας βέβαια θα πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη προσπάθεια για βιώσιμη επιχειρηματικότητα και βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Εξού και ήταν σημαντική η συνεργασία μας τα τελευταία χρόνια με τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη για νέες πρωτοβουλίες ε, σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική πολιτική. Δεν έχουμε ολοκληρώσει, έπονται και άλλες προτάσεις. Θέλουμε να έχουμε ένα ανθρώπινο κεφάλαιο για τις πρωτοβουλίες ε, της βιομηχανικής πολιτικής και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει και αηφορία στην ανάπτυξη στις θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε στην πρόθεση της επιχειρηματικότητας. Στα τελευταία χρόνια είχαμε την αρχική φάση της λειτουργίας ε, του μηχανισμού μικροπιστώσεων και επίσης στη νέα περίοδο χρηματοδότησης το πρόγραμμα για την απασχόληση και την ε, κοινωνική καινοτομία θα έχει επαρκή χρηματοδότηση για να στηρίξει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι και αυτό μια πηγή χρηματοδότησης πολλών προγραμμάτων για αναβάθμιση δεξιοτήτων, και επίσης για τη στήριξη, παραδείγματος χάρη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μεταξύ Είναι ένα θέμα Σημαντικό για την Ιταλία ή άλλες χώρες του Νότου της Ευρώπης. Επίσης, είμαι γνώμων προς ε, τον Γάλλο ε, που μίλησε για τον πίνακα επιδόσεων που πρόσφατα προτείναμε. Ελπίζω να λειτουργήσει καλά το εργαλείο αυτό και να συμβάλλει και στις συστάσεις αναχώρια για την προσεχή περίοδο. Τώρα, κατά πόσο χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία και τελειοποίηση, αυτό θα το δούμε σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Ωστόσο, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μια πρόσθετη ανάλυση σε αυτό το πίνακα επιδόσεως, σε αυτό το scoreboard, που καλύπτει ένα ευρύτερο πλαίσιο και άλλους δείκτες, πλέον ε, των πέντε αυτών βασικών δικτών. Ο Λιρέν αναφέρθηκε ήδη στο θέμα των ε, συντάξεων στην Ολλανδία. Να προσθέσω απλά ότι το 2012 ήταν ε, παραγωγική χρονιά για την ενεργό γύρανση και τη γυναική αλληλεγγύη. Πολλές θετικές δράσεις ε, προβλήθηκαν, οι οποίες καταδεικνύουν ότι μπορεί κανείς να εργάζεται περισσότερο, για περισσότερα χρόνια, εφόσον και οι γυναίκες και οι άνδρες σε πολλές χώρες ζουν περισσότερα χρόνια και η σύνδεση της, ε, του ορίου ε, συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Όμως, ε, πριν από δύο χρόνια, εγκρίναμε μια λευκή βίβλο για τις συντάξεις. Με πολύ καλή συνεισφορά και από την Ολλανδία, στην παρόδο. Πρέπει να σας πω ότι τώρα εκπονούμε, μάλλον προετοιμάζουμε μια συνεδρίαση, ένα συνέδριο για τις επόμενες εβδομάδες εδώ στις Βρυξέλλες που θα κάνει ένα απολογισμό της υλοποίηση αυτής της Λευκής Βίβλου. Θα συζητηθούν θέματα όπως ε, η φορητότητα των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων ή οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συντάξεων που έχουν ε, εφαρμοστεί από πολλά κράτη-μέλη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, θα υποβληθούν και θα παρουσιαστούν καλά μοντέλα, καλά μέτρα, τα οποία ελπίζουν να αποτελέσουν και έμπνευση για άλλες χώρες που ενδεχομένως υπολείπονται στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κ. Έκης από την Ουγγαρία, και θα απαντήσω στα ουγγρικά, επειδή ανέφερε κάποια πράγματα ε, ο βουλευτής αυτός, πραγματικά πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τη μακροοικονομική σταθερότητα στην Ουγγαρία. Παρακολουθούμε πάρα πολύ την κατάσταση. Εμείς προτείναμε η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος να κλείσει και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Φαίνεται η διαδικασία αυτή του ελλείμματος να έχει στεφθεί με επιτυχία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απασχόληση, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε μια βελτίωση. Πέραν των στατιστικών στοιχείων όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα είναι η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού. εντάθηκε, εντάθηκε συγγνώμη, τα τελευταία χρόνια στην Ουγγαρία. Επίσης ενισχύθηκαν οι δημόσιες υπηρεσίες. Δεν πρέπει να μας ε, διαφεύγουν αυτοί οι οι νέοι παράγοντες που ε, αναδύονται. Ξέρετε ότι σε περίοδο κρίσης αυξάνονται οι δημόσιοι πάλι. Είναι μια τάση αυτή. Αλλά αυτό δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να βρεθεί διέξοδος από την κατάσταση αυτή. Δηλαδή πώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει θέσεις εργασίας χωρίς απλά να δημιουργεί θέσεις στο δημόσιο τομέα. Δεν είναι αυτό η πιο ε, κατάλληλη μορφή αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού. Επίση, ε, τονίστηκε πάρα πολύ η σημασία τη εκπαίδευση και κατάρτιση. Για μα είναι θετικό αυτό, είναι σημαντικό στοιχείο. Και πρέπει να σα πω ότι ναι, πράγματι κατά το παρελθόν είχαμε ελλείψει, είχαμε αδυναμίε στην χρήση και αξιοποίηση των κονδυλίων, των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταία και η Κομισιόν και οι Ουγγρικές Αρχές εργάστηκαν εντατικά για την καλή αξιοποίηση αυτών των πόρων για να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι έγιναν όλα. Όχι. Ξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για σκληρή δουλειά και φέτος, γιατί έχουν μείνει πολλά εκκρεμή ζητήματα για το 2014. Όμως είναι Βέβαια ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε θετικά την πολύ σκληρή δουλειά της Ουγγαρίας. Μειώθηκε η διασπάθηση των πόρων στην Ουγγαρία. Απομακρύνθηκε η απειλή της κρίσης που πλανά το επάνω από την Ουγγαρία τους τελευταίους μήνες. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει να κλείσει ο εισηγητής. Όχι. Ωραία. Λοιπόν. We can conclude. Μπορούμε να κλείσουμε. Ευχαριστούμε τους επιτρόπους και όλους σας, εξ ονόματος και του Συμπρόεδρου κ. Δερμετζόπουλο, να σας θυμίσω ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο δείπνο στις 7 από διοργανώνει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σούλτς και ο πρόεδρος ε, του Ευρω... της Ελληνικής Βουλής ο κ. Ευαγγέλος Μαράκη θα τα πούμε σε λίγο εκεί. Oi oi, oi.